Λοιπόν, αγαπητοί συνάδελφοι, καλώς ορίσατε θερμά. Συνεχίζεται η συνεδρίαση της Επιτροπής μας. Συζητήσαμε χτες, συζητήσαμε σήμερα το πρωί και ερχόμαστε στην απογευματινή συνεδρίαση. Ξέρετε ότι αναβάλαμε το σημείο 10, δεν θα συζητηθεί, το είπαμε από χτες αυτό. 11 και 12 είναι η ασφάλεια του εφοδιασμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε φυσικό αέριο θα θέλαμε να χωρίσουμε αυτά τα δύο θέματα. Τι εννοώ. Να ασχοληθούμε πρώτα με την εκτίμηση αντικτύπου, να ενημερωθούμε και να κάνουμε και ερωτήσεις, διότι καμιά φορά σε προηγούμενες συζητήσεις είχαμε ε, το φαινόμενο να μην ε, ασχοληθούμε γιατί δεν είχαμε χρόνο με τα θέματα του αντικτύπου και της μελέτης αντικτύπου αν υπάρχουν ερωτήσεις, δηλαδή αν υπάρχουν συμπληρωματικές ερωτήσεις, διευκρινιστικές, ε, αν συμφωνούμε ή όχι. Και από εκεί και πέρα να συζητήσουμε την πολύ συγκεκριμένη πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Καλώς ορίζω από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή τον κύριο Γενικό Διευθυντή της Γενικής Διεύθυνσης ε, Μεταφορών και Ενέργειας, τον κύριο ε, Ρούιτε και τον κύριο Βιλμέ, τμήματάρχη. Και συμφωνήσαμε κύριο Ρούιτε να πει κάποια εισαγωγικά και μετά να ακούσουμε τα θέματα της μελέτης αντικτύπου και του κανονισμού. Έχετε το λόγο κύριε Ρούτσε, παρακαλώ. Καλώς όριστε θέρμα. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θα μιλήσω αγγλικά. Αν μου επιτρέπετε. Βεβαίως αν θέλετε μετά απαντάω και στα γερμανικά. Θα σας κάνω μια σύντομη εισαγωγή για το τι κάναμε ως προς τον κανονισμό για την ασφάλεια εφοδιασμού σε φυσικό αέριο. Ξεκινώντας με τα πολιτικά, πιο καλή αξιολόγηση επιπτώσεων για την ασφάλεια σε αέριο ήταν η κρίση Ρωσία-Ουκρανία για το αέριο στις αρχές του 2009 όπου κάπως καταφέραμε σε όλα τα επίπεδα να έχουμε καλή συνεργασία. αλλά σε νομικό κενό. Συνεργασία εταιριών, συνεργασία κρατών μελών και περιφερειακά και συνεργασία εταιριών, κρατών μελών και της Κομισιόν. Σας είπα σε νομικό κενό. Διότι χρειάστηκε να πάρουμε αποφάσεις και να χρησιμοποιήσουμε εργαλεία που δεν έχουν νομική βάση. Όπως η τοποθέτηση, η υποστολή και η τοποθέτηση παρατηρητών στην Ουκρανία πολύ στενή συνεργασία ακόμα και σε επίπεδο πρωθυπουργών και έτσι επιταχύναμε την πρόταση για τον κανονισμό για την ασφάλεια όσον αφορά το αέριο και κάναμε και μία λεπτομερή εξέταση αξιολόγηση των επιπτώσεων. Από την εμπειρία μου σας λέω ότι όσο πιο καλή είναι αυτή η αξιολόγηση, τόσο πιο καλή είναι η διαδικασία λήψης των αποφάσεων. Γιατί έχουμε τα νούμερα, έχουμε τα δεδομένα, τα μελετάμε, τα συζητάμε και μετά η διαδικασία λήψης των αποφάσεων έτσι επιταχύνεται. Σας προτείνω εγώ και συνάδελφός μου να σας πούμε δύο λόγια για την ε, αξιολόγηση επιπτώσεων μετά στη διάθεσή σας για ερωτήσεις και μετά θα σας παρουσιάσουμε τον κανονισμό. Παρακαλώ Επιτρέψτε να μιλήσει ο συνάδελφος. Ο κύριος Σουρίτε. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Ας δούμε γρήγορα την αξιολόγηση επιπτώσεων. Μέσα στα πλαίσια της γενικής κρίσης δεν πιο καλή αξιολόγηση μπορούσαμε να κάνουμε. Τον Ιανουάριο είχαμε την κρίση που μας έδειξε τι μπορεί να σημαίνει αν υπάρξει μια διακοπή παροχής στην Ουκρανία για την Ένωση. Και είχαμε αντιδράσεις σε όλη την Ένωση που πρέπει να τις μελετήσουμε διότι βάσει αυτής εδώ της αξιολόγησης σε μεγάλο βαθμό η βάση επηρεάζεται από το τι έγινε τον Ιανουάριο. Το Ηνωμένο Βασίλειο που δεν υπέστη άμεση διακοπή του ρωσικού αερίου έστειλε αέριο προς την Ευρωπαϊκή Ήπειρο για να διευκολύνει αυτή τη διακοπή που συνέβη στην Ουκρανία. Στην πραγματικότητα λοιπόν μια διακοπή επηρεάζει όλη την Ένωση που είναι εσωτερική αγορά. Είδαμε επίσης ότι η διακοπή μέσα στην Ένωση επηρέασε 12 χώρες μέλη και πολλές άλλες χώρες των Δυτικών Βαλκανίων. Άλλες με διακοπή 100% άλλες με 20%. Όσο πιο μακρά ήταν από την Ουκρανία η κάθε χώρα, τόσο πιο ήπια η επίπτωση. Αλλά και Ευρωπαϊκέ χώρες υπέστησαν δεινό πλήγμα. Διοκοπή δύο εβδομάδων στον αγωγό Μέσο Ουκρανίας και είδαμε τι πάει καλά γιατί δεν πάει καλά. Είδαμε ότι ορισμένα λειτουργήσαν. Παραδείγματο χάρη η εσωτερική αγορά είναι καλό εργαλείο για την ασφάλεια. Επίσης είδαμε ότι οι εταιρείε ήταν σε θέση να συμφωνήσουν βραχυπρόθεσμα για παροχή την τελευταία στιγμή ορισμένες χώρες που είχαν μεγάλη ανάγκη. Ορισμένες χώρες ήταν καλά προετοιμασμένες είχαν επαρκή προγράμματα έκτακτης ανάγκης. Είδαμε μια ομάδα συντονισμού για το αέριο της Ένωσης να συντονίζεται και με τους εκπρόσωπους της βιομηχανίας και με τις χώρες μέλη. Η Κομισιόν συνεργάστηκε με την ομάδα αυτή. Είπα δεν πει στο όφελος της αντίστροφης ροής. Δηλαδή πολλοί αγωγοί λειτουργήσαν αντίστροφα από τη Δύση προς την Ανατολή. Λειτουργήσε αυτό. Το είδαμε σε δύο περιπτώσεις. Βουλγαρία, Ελλάδα, Τσεχία, Σλοβακία. Πολύ σημαντικό αυτό, πολύ σημαντικό δίδαγμα. Τέλος, όλα τα νοικοκυριά παρέμεινε εφοδιασμένα με εξαίρεση τη Βουλγαρία που υπέστη το πιο δεινό πλήγμα. Αλλά και ορισμένα πράγματα δεν πήγαν καλά, όπως ελλείψεις υποδομών, το να φτάσει στο έργο εκεί που το χρειάζονται. Αυτό ήταν η κύρια αιτία των σοβαρών συνεπειών. Μερικές χώρες δεν ήταν καλά προετοιμασμένες για την κρίση και πλήρωσαν το τίμημα. Η ανταλλαγή πληροφοριών και η διαφάνεια δεν ήταν πάντα επαρκής. δεν υπήρξε επαρκής συντονισμός διασυνοριακά για τα έκτακτα μέτρα. Είδαμε ε, αρνητικά εθνικά μέτρα που επηρέασαν άλλες χώρες, μονόπλευρα μέτρα δηλαδή, που προξένησαν ζημιά σε γειτονικέ χώρες. Είδαμε πίσω ότι δεν υπάρχει αλληλεγγύη μεταξύ των κρατών μελών δεν υπήρχαν συμφωνίες μεταξύ των κρατών μέλων για αλληλοβοήθεια και είδαμε ότι μερικές φορές υπήρξε επαρκής αξιολόγηση των κινδύνων. Αυτά για την κρίση του Ιανουαρίου. Η Κομισιόν για να προετοιμάσει αυτό τον κανονισμό και να κάνει την αξιολόγηση στηρίχτηκε σε όλε αυτές τις παρατηρήσεις του Ιανουαρίου. συζητήσουμε με όλους τους ενδιαφερόμενους, κρατημέλη, κομισιόν, να δούμε τι ακριβώς συνέβη. Και έχουμε πέντε επιλογές. Πρώτον, να μην έχουμε νέα μέτρα, status quo δηλαδή. Το δεύτερο, καλύτερη εφαρμογή της Οδηγίας 2004-67. Τρίτη, ε, μια οικούσια η προαιρετική προσέγγιση μέσα βιομηχανία. τέταρτο μια αναθεώρηση τη οδηγίας 2004-67 και τέσσερα ρύθμιση όσον αφορά την ασφάλεια για το αέριο. Ας πάρουμε το πρώτο. Να μην ληφθούν μέτρα σε επίπεδο ένωσης. Αυτό αστηρίζεται στο τρίτο πακέτο της εσωτερικής αγοράς του Ιουνίου Δούμε τι προβλέπει το οικονομικό πρόγραμμα ανάκαμψη, ιδιαίτερα όσον αφορά την υποδομή και μελλοντική αναθεώρηση όπως έχει προβλεφθεί για το 2010. Αλλά αυτή η αξιολόγηση αυτή τη λύση μας οδήγησε στο συμπέρασμα ότι δεν είναι υπεύθυνη όσον αφορά την ασφάλεια. Δεν έχουμε πρότυπα προδιαγραφές για να αξιολογήσουμε ασφάλεια και δεν υπάρχουν και κίνητρα για επενδύσει για την υποδομή που απαιτείται. Επίσης δεν υπάρχουν και ειδικέ διατάξεις για συντονισμό σε έκτακτη ανάγκη και ούτε μηχανισμός αγιλεγγύης. Αυτή η λύση δεν τη θεωρήσαμε ότι υπόσχεται πολλά. Δεύτερη λύση. Καλύτερη εφαρμογή της οδηγίας 2004-67. Κάναμε έκθεση για την εφαρμογή αυτής της οδηγίας. Δημοσιεύτηκε και αυτή ταυτόχρονα με τον κανονισμό τον Ιούλιο. Η οδηγία αυτή οδήγησε σε τεράστιες διαφορές στις προδιαγραφές που εφαρμόζονται από τα 20 κράτη-μέλη. Μόνο 10 κράτη-μέλη έχουν έκτακτα μέτρα συστηματικά με εθνικό πρόγραμμα. Δεν απαιτείται συντονισμός στην οδηγία και ο ορισμός δεν είναι σαφής όσον αφορά το ρόλο και την ευθύνη των διαφόρων φορέων και επίσης ε, οι απαιτήσει για αναφορά σε θέματα κρίσεως είναι ανεπαρκείς. Θεωρήσαμε λοιπόν ότι ακόμη και με διαδικασίες παράβασης όσον αφορά την οδηγία αυτή πάλι δεν θα πετυχαίναμε αυτό που θα θέλαμε. Περνάμε στην τρίτη λύση προαιρετική δράση εκ μέρους της βιομηχανίας. Είναι αλήθεια ότι ο κλάδος αυτός όταν μπει σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης οι φορείς της αγοράς είναι αυτοί που τροφοδοτούν την αγορά είτε αυτοί που μεταφέρουν είτε αυτοί που παρέχουν το αέριο ο ρόλος της είναι λοιπόν μεγάλος το θέμα είναι μπορούμε να στηριχτούμε μόνο σε αυτούς, στη δική τους δράση. Ξέρουμε ότι τα TSO συνεργάζονται και οι μεταφορείς με θελάσσια φορτία και αυτοί είναι σε θέση να κλείσουν βραχυπρόθεσμα συμβόλαια για να βοηθήσουν. Οι ρυθμιστές επίσης όπου υπάρχουν βοηθάνε και υπάρχει μια πρωτοβουλία της βιομηχανίας αερίου Βερολίνο Ιούνιος 2009 για την ασφάλεια. Αλλά αυτό δεν οδηγεί κατά ανάγκη σε μια ενιαία μέθοδο για την ασφάλεια εφοδιασμού, διότι δεν υπάρχουν κοινέ προδιαγραφές που είναι σημαντικός, προκειμένου να υπάρχει ευθύνη και αγγελική και η ασφάλεια εφοδιασμού τελικά ως θέμα, είναι ένα θέμα δημόσιας τάξης έχει σχέση με την ε, ευθύνη της κάθε χώρας. Φερεπίν, η Γαλλία ξέρει ότι η ασφάλεια εφοδιασμού είναι ένα βασιλικό προνόμιο κατά κάποιο τρόπο. Δηλαδή ουσιαστικά ανήκει στην αποκλειστική ευθύνη του κράτους. Μόνο να στηριχτούμε λοιπόν στη βιομηχανία δεν αρκεί. Πρέπει όλοι να συνεργαστούν. Περνάμε στην τέταρτη λύση. Αναθεώρηση της οδηγίας 2004. Έχουμε δείξει ότι πρέπει να αναθεωρηθεί αυτή η οδηγία με την έκθεση για την εφαρμογή της 2004 του 67. Επίσης υπάρχει ανάγκη να προσαρμογεί το πλαίσιο στο νέο ρυθμιστικό πλαίσιο που δημιουργήθηκε με το τρίτο πακέτο εσωτερικής αγοράς. Αλλά αυτό που διαπιστώσαμε, ειδικά για τη βιομηχανία τώρα, είναι ότι η βιομηχανία θα έπρεπε να παίρνει πλήρες μέρος στη διαδικασία αυτή. Είναι οδηγία αφορά μόνο τα κράτη-μέλη. Χρειάζεται μακρός χρόνος μεταγραφής της οδηγίας στην εθνική νομοθεσία. Αυτό θα οδηγήσει σε μεγάλες διαφορές μεταξύ των κρατομελών και το είδαμε αυτό. Και δεν θα οδηγήσει σε εμπιστοσύνη και αλληλεγγύη που απαιτείται να υπάρχει στο σύστημα για να αντιμετωπίσουμε έκτακτες ανάγκες. Και έχουμε και διαφορετικές προδιαγραφές σε κάθε χώρα, οπότε δεν δημιουργείται ε, συνθήκες ε, ε, ανταγωνισμού ίσο για όλους. Και περνάμε στην επόμενη λύση. Η ρύθμιση της ασφάλειας όσον αφορά την παροχή αερίων. Είδαμε ότι αυτό δίνει σαφήνεια και ακολουθία όσον αφορά τις προδιαγραφές και τις υποχρεώσεις όλη την Ευρώπη. Και έτσι εξασφαλίζεται αλληλεγγύη. Είδαμε ότι ε, σε ένα ρεαλιστικό σενάριο διακοπής της, του εφοδιασμού που έγινε το Ιανουάριο απαιτείται, απαιτούνται συγκεκριμένες προδιαγραφές για υποδομή, για την παροχή, ενέδωσε εναρμόνιση ο κανονισμός θα εφαρμόζεται άμεσα για όλους. Δημόσιες αρχές, αυτοί που παρέχουν το αέριο, αυτοί που μεταφέρουν το αέριο, μια καλή βάση συνεργασίας. Επίσης, σαφώς ορίζεται η εμπλοκή θετικά της Κομισιόν και δεν χρειάζεται για πολλή χρόνος για να μεταγραφεί το κείμενο αυτό στην Εθνική Νομοθεσία. Αυτές ήταν οι πέντε επιλογές που μελετήσαμε που επηρεάζονται, όπως σας είπα, από τα διδάγματα του Ιανουαριού. Γι' αυτό υπάρχει ένα κείμενο που διηγείται την ιστορία αυτή του Ιανουαρίου και το τι διδάγματα αντλούμε. Θα σταματήσω εδώ κύριε Πρόεδρε για να επιτρέψω να περάσουμε στην χρόνο να περάσουμε στη συζήτηση. Ευχαριστώ πολύ. Ακούσαμε λοιπόν τις εξηγήσεις, την παρουσίαση της μελέτης αντικτύπου. Τώρα έχετε και εσείς την ευκαιρία να κάνετε ερωτήσεις επάνω σε αυτό, έτσι, για τη μελέτη αντικτύπου και επιπτώσεων. Αν χρειάζονται διευκρινήσεις κάποια σημεία ή αν θεωρείτε ότι πρέπει να ακούσουμε κι άλλα σε πρώτη φάση νομίζω καλό θα ήταν να τα συζητήσουμε. Ο συνάδελφο Βιντάλ Κουάδρα ζήτησε πρώτο το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ και τον κύριο Γενικό και τον κύριο Διευθυντή για την παρουσίαση αυτή της μελέτης αντικτύπου για την νομοθεσία αυτή, για την ασφάλεια στην προμήθεια φυσικού αερίου. Μια γενική εντύπωση που αποκομίζει κανείς ακούγοντάς σας. Γιατί διαβάζοντα προσεκτικά και μελετώντας το έγγραφο είναι ότι ο κανονισμός που αρχίζουμε σήμερα συζητάμε ήταν απολύτως απαραίτητος. Δηλαδή είναι ένα νομοθέτημα το οποίο δεν είναι καρπός μιας ε, αυθόρμητης έμπνευσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αλλά απαντάει σε μια πραγματική ανάγκη. Από εκεί και πέρα τώρα, χωρίς καμία αμφιβολία, η μελέτη αντικτύπου μπαίνει σε πολλά συγκεκριμένα θέματα. Και κάτι που θα με ενδιαφέρει εμένα είναι το εξής. Το Συμβούλιο, το οποίο σε τελική ανάλυση είναι ο εταίρος μας σε αυτή την υπόθεση, η εκπόνηση της νομοθεσίας εξέφρασε κάποιες ε, ανησυχίες και δεν ξέρω αυτό θα παίξει στη συναπόφαση. Τη μελέτη αυτή του αντικτύπου γίνονται και ποσοτικές εκτιμήσεις ε, σχετικά με το κόστος, έτσι. της εφαρμογής του τύπου νη μείον ένα στα διάφορα κράτη-μέλη. Και επειδή η γλώσσα της μελέτης αυτής αντικτύπου είναι συγκρατημένη και νυφάλαια κάπως, ε, συνάγει κανείς από τις επιπτώσεις και από τις εκτιμήσεις, όταν τα διαβάζει όλα αυτά, ότι όταν τεθεί σε ισχύ ο κανονισμός για να καλυφθούν όλες αυτές οι διατάξεις, το κόστος στα διάφορα κράτη-μέλη δεν θα είναι καθόλου ομοιόμορφο σε καμία περίπτωση. Δηλαδή θα έχουμε κράτη-μέλη όπου το κόστος προσαρμογής θα είναι πολύ υψηλό και άλλα κράτη-μέλη που θα είναι πολύ πιο βατό. Ερωτώ λοιπόν, μέχρι ποιο βαθμό η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πιστεύει με τα στοιχεία αυτά τα αριθμητικά αυτή η ετερογένεια του κόστους και οι αποκλήσει στα κράτη-μέλη, όταν λέω τεθεί σε ισχύ ο νέο κανονισμό, τι πιστεύει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αυτό νομίζετε εσείς ότι θα δυσκολέψει την έγκρισή του. Και τι είδους μηχανισμοί προβλέπονται αλληλεγγύης, χρηματοδότησης, για να ξεπεραστούν, να διασκεδαστούν οι επιφυλάξει ορισμένων κρατών μελών που πλήττονται ιδιαίτερα από το κόστος. Ευχαριστώ. Ε, αν θέλετε να απαντώνετε κατευθείαν ερωτήσει, είναι πιο έξυπνο, γιατί είναι πάρα πολύ στεναρέ και αποφασιστικές. Κύριε κύριος παρακαλώ. Ε, Ευχαρίστω. Θα ήθελα να σχολιάσω και την αξιολόγηση του δικτυ νη 1 και τις εκτιμήσεις κόστους, οι οποίες περιλαμβάνονται σε έναν πίνακα. Αυτός ο πίνακας ε, δείχνει περίπου τα, τις διαφορετικές δαπάνες ε, για τα κράτη-μέλη με τη εισαγωγή του νέου προτύπου. Είναι ένα ταμπλό, ένα πίνακα, στον οποίο έχουμε in τι, θα κοστίσουν οι αλλαγές που θα γίνουν και βλέπουμε ότι τις τελευταίες, ε, τους τελευταίους μήνες ε, που έχουμε ασχοληθεί με το σύστημα οικονομικής ανάκαμψης ε, το, το πρότυπο νη μείον ένα θα μπορέσει να το, να, θα μπορέσουμε να το εφαρμόσουμε σε ορισμένα κράτη-μέλη εκεί όπου έχουν προβλεφθεί τέτοια, προβλήμα, τέτοια έργα, τέτοια προγράμματα ε, ανάκαμψης, οικονομικής ανάκαμψης. Δεύτερη παρατήρηση. Στην, στον κανονισμό προβλέπεται ε, μία περιφερειακή συνεργασία. Όσο περισσότερο συνεργαζόμαστε περιφερειακά, τόσο χαμηλώνει το κόστος. Εάν ένα κράτο θέλει μόνο του να επιτύχει το πρότυπο νήμιον 1, το δίκτυο νήμιον 1, τότε μπορεί να το επιτύχει, ε, αλλά μπορούν, και δύο κράτη-μέλη να συνεργαστούν, όπως η Βουλγαρία και η Ελλάδα, διότι έτσι θα αποφυληθούν από, την, ε, ε, από τα αλληλοσυμπληρούμενα στοιχεία της, υποδομής. Είναι όμως δύσκολο τον προτέρων να καθορίσουμε ακριβώ το κόστος, διότι μπορεί μεμονωμένα να ακολουθήσει την πορεία των κράτων μέλο ή μια συνδυασμένη πορεία κρατών μελών. Για, γι' αυτό είναι δύσκολη η αξιολόγηση του δικτυνή μείον ένα. Ευχαριστώ κύριε Τσιμάνσκι. Ευχαριστώ. Ο κανονισμός επιτρέπει δύο χρόνια για την ε, ολοκλήρωση της ε, αντίστροφης ροής ε, των σημερινών ροών φυσικού αερίου. Δεν νομίζω ότι φτάνει αυτός ο χρόνος, δεδομένου ότι αυτές οι επενδύσεις θα πρέπει να έχουν και μια οικονομική αιτιολόγηση και εδώ μιλάμε για τεράστια ποσά. Τώρα, τι κατάσταση επικρατεί όσον αφορά τι κρατικέ ενισχύσει. Οι κρατικέ ενισχύσει θα τι αντιμετωπίσουμε διαφορετικά σε αυτό το προϊόν, σε αυτό τον τομέα, από ότι ε, σε άλλου τομεί. Θα αντιμετωπιστούν διαφορετικά λοιπόν σε αυτόν τον κανονισμό. Οι ενδιαφερόμενοι, οι οποίοι ας πούμε θα ζημιωθούν, θα χάσουν χρήματα, θα αποζημιωθούν από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν νομίζω ότι μία αποζημίωση ε, βασιζόμενη σε συγκεκριμένες ε, ταρίφες ε, είναι δυνατόν να, να δοθούν στην αγορά φυσικού αερίου έχουμε ιδιαιτερότητες και πρέπει να λάβουμε υπόψη αυτές τις ιδιαιτερότητες ως επίγουσες διότι δεν πρόκειται μόνο να υποφέρει ή μια, να υπάρχουν επιπτώσεις πάνω σε μια χώρα, αλλά μια λυσίδα χωρών. Και επίσης 7 μέρες νομίζω δεν φτάνει για να γίνει μία ανακοίνωση κατάστασης έκτακτης ανάγκης αυτή η 7 περίοδος. Πιστεύω ότι ο κανονισμός πρέπει να εξετάσει και τα, το θεμελιώδε θέμα των εξω, της εξωτερικής προμήθειας φυσικού αερίου. Αυτό είναι πολύ κρίσιμο για, την, τον εφοδιασμό. Ε, πέραν δηλαδή από την διακρατική, διευρωπαϊκή και την εξωτερική. Ευχαριστώ, ε, λέει ο πρόεδρος. Θα συζητήσουμε μόνο αυτή την έκθεση αξιολόγηση επιπτώσεων και μετά τα υπόλοιπα. Ε, εντάξει, όχι ότι έχουμε ξεχωρίσει ε, το θέμα αυτό ε, στο παρελθόν, αλλά το συζητήσουμε τώρα μεμονωμένα, έτσι, μόνο αυτό το θέμα. Ε, εάν μου επιτρέπετε, θα προσπαθήσω να απαντήσω, λέει ο η δυνατότητα αντίστροφης ροής των αγωγών και οι μελέτες που έχουν γίνει δείχνουν ότι το κόστος θα είναι χαμηλότερο από ό,τι τελικά νομίζαμε. Το κόστος ε, διαφέρει, κυμαίνεται από 1 έως 5 εκατομμύρια ανάλογα με το τι δυναμικό ροής προβλέπεται. Στο πρόγραμμα οικονομικής ανάκαμψης έχουμε και μία προβλέψη, μία πολύ μεγάλη εγκατάσταση 80 εκατομμυρίων για αντίστροφη ροή. Αυτά θα είναι φρέσκα ευρωπαϊκά κονδύλια για την αντίστροφη δυναμικότητα ροής, για το αντίστροφο δυναμικό ροής. Ο, τώρα πώς, πότε θα μπορέσουμε να εκμεταλλευτούμε αυτή την αντίστροφη ροή, πότε έχει νόημα μέσα στο πλαίσιο της ασφάλειας του εφοδιασμού, ας πούμε από την ε, Ανατολική Πολωνία προς Ανατολάς. Ε, έτσι όπως έχουμε διατυπώσει αυτό το σκέλος της ε, αντίστροφης ροής στον κανονισμό, προσφέρουμε τη δυνατότητα να πει κάποιος ότι δεν χρειαζόμαστε, δεν χρειάζεται αυτή η αντίστροφη ροή και μέσα στη διαδικασία που και, μελέτη ε, αυτό, αυτής της ε, πρότασης θα, καθορίσουμε εάν η σχέση αυτή η κόστους ωφέλους είναι σωστή ή όχι. Θα το μελετήσουμε. Όταν, όσον αφορά τις κρατικές ενισχύσεις για την αντίστροφη ροή, δεδομένου ότι η επάρκεια εφοδιασμού είναι κρατική μέρη, μια κρατική ευθύνη θα ισχύσουν ε, οι ήδη κανονισμοί όπως σε μια κρατική επιχείρηση, δημόσια επιχείρηση. Όμως έχουμε προβλέψει και στον κανονισμό ότι οι δαπάνες των εγκαταστάσεων αντίστροφης ροής μπορούν να ενσωματωθούν μέσα στη... I the στα τιμολόγια. Και πολλά, πολλές ε, ερωτήσεις έχουν ήδη απαντηθεί από το άρθρο 6, παράγραφος 5 του κανονισμού. Ε, διαισθάνομαι ότι υπάρχουν πολλές ακόμα απορίες πάνω σε αυτό το θέμα, οι οποίες όμως θα απαντηθούν κατά την πρόοδο των διαπραγματεύσεων για τον κανονισμό. Ευχαριστώ κύριε Σβόμποντα. Ευχαριστώ. Μία ερώτηση έχω μόνο. Είπατε ότι υπάρχει σχέση μεταξύ του recovery προγράμματος ανάπτυξης και άλλων ε, ε, προτάσεων του κανονισμού ε, και επιπτώσεων που θα έχει ο κανονισμός. Ο κανονισμός. Ορισμένες επιπτώσεις θα μειωθούν σε σημασία βεβαίως εφόσον αναπτυχθεί το, πρόγραμμα ανάπτυξης στο πρόγραμμα οικονομική οικονομικής ανάκαμψης. Έχουμε συζητήσει το θέμα αυτό ε, με την Κομισιόν στο παρελθόν και σήμερα το πρωί η Επίτροπο κυρία Ρέντινγκ μα είπε ότι δεν είναι καθόλου ευχαριστημένη για την ε, χρησιμοποίηση των πόρων από πλευρά κρατών μελών. Δεν ξέρω, ίσω στον τομέα της ενέργεια ε, η χρήση, η απορρόφηση και χρήση των πόρων να είναι καταπληκτική, εξαιρετική και εσεί να μα πείτε καλύτερα νέα πώς κρίνει η Κομισιόν τη δραστηριότητα των κρατών μελών, το τι έχουν κάνει δηλαδή μέχρι τώρα για το, πρόβλημα, για το θέμα της οικονομικής ανάκαμψης. Ευχαριστημένοι ή όχι. Ε, δεν είμαι σε θέση εδώ ακριβώς να σας <clears throat> παρουσιάσω τα αποτελέσματα, τα συμπεράσματα μη αξιολόγηση η οποία ακόμα εξελίσσεται. Αλλά υπολόγισε ότι πάνω από 70% των ε, πιστώσεων μπορεί να δαπανηθεί γρήγορα και είμαι βέβαιος ε, ότι θα κερδίσω το στοίχημα. Ε, μία πρόταση ήταν όλη αυτή. ναι, μία πρόταση, μία ενέργεια. Μία πρόβλεψη. έχουμε προχωρήσει αρκετά στην αξιολόγηση και κατά βάση η σκληρή δουλειά που έκαναν όλοι οι συνεργάτες ε, κατά το καλοκαίρι έχει δώσει αποτελέσματα θετικά. Πολύ ωραία λέει ο Πρόεδρος. Περιμένουμε λοιπόν τους τελικούς, τα τελικά στοιχεία. Ο κύριος Μπρεζίνα. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω, Κομισιόν, για την πρότασή σας, για τον κανονισμό. Είναι πάρα πολύ χρήσιμη πρόταση. Τώρα απαιτείται να ακολουθεί μία προτεραιότητα, το κριτήριο ασφάλειας νημείων 1. Και δεν πρέπει να υποχωρήσουμε σε καμία περίπτωση ούτε να ε, μετριάσουμε την δύναμη αυτής της απόφασης. Μιλάμε για το κόστος της απόφασης νήμιον 1 και η ερώτηση μου είναι τι μηχανισμοί μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να βοηθηθούν χώρες που έχουν τα πιο μεγάλο έγκυμα όσον αφορά το νήμιον 1. Ξέρω ότι η ερώτηση αυτή είναι πολύ λεπτή γιατί μπορεί να μπούμε στον πειρασμό να παίξουμε κατά κάποιο τρόπο με τις δυνάμεις της αγοράς. Η ερώτησή μου προς την Κομισιόν είναι, θεωρείτε ότι αυτός ο κανονισμός που προτείνεται επαρκεί για να αντιμετωπιστεί η επόμενη παρόμοια κρίση, παρόμοια όπως αυτή του Ιανουαρίου. Ξέρω ότι το θέμα αυτό είναι πάρα πάρα πολύ λεπτό. δεν έχουμε μια ενεργειακή πολιτική. Η ενεργειακή πολιτική ακόμα είναι στα χέρια της κάθε κυβέρνησης. Υπάρχουν άλλα μέτρα που θα μπορούσαν να προταθούν προκειμένου να προλάβουμε μια επόμενη κρίση. Απάντηση. Κύριε Βρεζίνα, φυσικά ο κανονισμός είναι μόνο ένα στοιχείο μεταξύ πολλών άλλων. Δεν νομίζω ότι ο κανονισμός μόνος του λύνει τα πάντα. Είχα την ευχαρίστηση να παρακολουθώ τα θέματα αυτά από κοντά τα τελευταία τέσσερα χρόνια στον αφορά την ενεργειακή πολιτική. Στην αρχή λοιπόν, γύρω στο 2006 δηλαδή, είχαμε μια κρίση αερίου. Τότε συζητούσαμε με το Κοινοβούλιο τα ε, διευρωπαϊκά ενεργειακά δίκτυα και όλοι συμφωνούσαμε ότι τα δίκτυα αυτά θα πρέπει να χρηματοδοτηθούν ιδιωτικά 140 εκατομμύρια 7 χρόνια ότι επαρκούσαν για την υποδομή. Και τελικά όλοι είδαμε ότι αυτό δεν αποδείχθη αληθινό. Δηλαδή υπήρξαν περιπτώσεις, υπάρχουν περιπτώσεις όπου έχει νόημα να υπάρχει ιδιωτική χρηματοδότηση δικτύων. Και είμαι σίγουρο, γιατί ο πρόεδρος Μπαρόζο το έχει ήδη ανακοινώσει, θα γίνει μια συζήτηση του χρόνου για την ευρωπαϊκή πολιτική υποδομών για ενεργειακά δίκτυα και φυσικά η συζήτηση για τα διευρωπαϊκά ενεργειακά δίκτυα θα επηρεαστεί από το πρόβλημα ασφάλειας εφοδιασμού. Ας μην μπερδεύουμε αυτά τα δύο πράγματα. Να είμαστε υπέρ των υποδιαγραφών νήμιον 1. Ο κανονισμός δεν είναι ο κατάλληλο επίπεδο για να ε, φροντίσουμε να υπάρξουν περισσότερα κονδύλια. Πρόεδρος, ευχαριστούμε. Ο κύριος Βόγκανα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Όπως και τα περισσότερα μέλη εδώ του Κοινοβουλίου θεωρούν ότι είναι σημαντικό αυτό το θέμα και δεν μπορούμε να το αφήσουμε στα χέρια της αγοράς και μόνο. Και χαίρομαι για τον κανονισμό. Έχω ε, μια-δυο αμφιβολίες ή ανησυχίε. ανησυχίες. Το πρώτο, θα πρέπει να διευκρινίσουμε τις εξουσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής εκεί και των κρατών μελών όταν υπάρχει έκτακτη ανάγκη. Με άλλα λόγια, πότε θα έχουν ε, την εξουσία τα κράτη-μέλη και πότε θα επεμβαίνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Θα βάλετε στον κανονισμό καμία σχετική διάταξη για να ξέρουμε εκεί τι γίνεται. Ο I, um, want to underline that the... Θα ήθελα να τονίσω το εξής. Και ήδη όπως βλέπετε συζητάμε τον κανονισμό. Η πρότασή μας λοιπόν του κανονισμού λέει τα εξής. Πρώτον, ασφαλής ανεφοδιασμός στηρίζεται στην ιστορική αγορά. Δεύτερον, στηρίζεται σε προληπτικά μέτρα. Άρα, η ανάλυση των κινδύνων και η εφαρμογή υποδομής είναι πιο σημαντική από ότι η αντίδραση έκτακτης ανάγκης βέβαια από τη στιγμή που θα έχουμε την ανάλυση του κινδύνου τα μέτρα τα προγράμματα έκτακτης ανάγκης ίσως προσωρινά ή όχι θα πρέπει να υπάρχουν πολλά επίπεδα δράση και φυσικά θα ισχύσει και αρχή της επικορικότητας Πρώτη βιομηχανία μετά τα κρατημέλη ιδιωδώς σε συνεργασία και μόνο μετά κοινωτική δράση. Ορίζουμε σε ποιο χρόνο θα πρέπει να λάβει χώρα κοινωνική δράση. Άρθρο 10. ως αντίδραση σε έκτακτα μέτρα που ήδη έχουν κινητοποιηθεί στα κράτη-μέλη και σε πλαίσια περιφερειακής συνεργασίας. Αυτό λειτουργήσε τον Ιανουάριο. Όλοι δηλαδή οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να συνεργαστούν. Όπως λέμε και στο άρθρο 3 του κανονισμού. Όπου αναφέρονται όλοι οι αρμόδιοι φορείς εθνικές αρχές, η βιομηχανία, οι πελάτες, οι κομισιόν, ο καθένας στο ρόλο του. Ευχαριστώ. Έχω δύο ακόμα μιλητές και έβαλα και το δικό μου όνομα στον κατάλογο. Λοιπόν, για την έκθεση αξιολόγησης καταρχάς, όποιος θέλει να ρωτήσει, ο κύριος Σούζα Βάγνερ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Πάρα πολύ σύντομα θέλω να πω το εξή. Καταρχάς ευχαριστώ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την τόσο αξιόλογη και σαφή παρουσίαση του προβλήματος. Ε, κατά δεύτερο λόγο θα ήθελα να πω ότι εμένα μου φαίνεται ότι είναι αναπόφευκτο να προχωρήσουμε σε έγκριση κανονισμού. Και αν έχει ακόμα κανένας καμιά αφιβολία, όταν δεν ξέρουν κάποιες χώρες πώς να λύσουν ένα πρόβλημα, φτιάχνουν ένα νόμο. Ε, ε, κυκλοφορεί αυτό και ισχύει και είναι και κίνδυνος αυτός. Αλλά ε, το να έχουμε κανονισμό είναι πολύ πιο αποτελεσματικό από ότι η οδηγία, όπως είπατε, γιατί η οδηγία χρειάζεται από εκεί και πέρα μεταφορά στα διάφορα κρατημέλη πάρα πολύ περίπλοκη και είναι πολύ μακροσκελής η διαδικασία. Ταυτόχρονα όμως θα πρέπει να πούμε ότι ο κανονισμός αυτός και είναι η πρότασή μου ή το αίτημά μου θα πρέπει να έχει συνταχθεί με αρκετή ευελιξία για να ληφθεί υπόψη η τελείως διαφορετική κατάσταση του κάθε κράτους μέλους. Δεν είναι το ίδιο δηλαδή από πλευράς εξάρτησης η κατάσταση της Ισπανίας με τις χώρες που βρίσκονται πιο κοντά γεωγραφικά στην Ανατολική Ευρώπη. Εδώ έρχομαι λίγο να συμφωνήσω με την ανησυχία που άκουσα από τον κύριο Βιδάλ Κουάδρας. Γι' αυτό λοιπόν ναι στον κανονισμό, αλλά ευέλικτο κανονισμό που να λαμβάνει υπόψη τις πολύ διαφορετικές απαιτήσει των ε, κρατών μελών. Ευχαριστώ. Εάν ε, μου επιτρέπετε πολύ γρήγορα να κάνω μια παρατήρηση Πραγματικά χρειαζόμαστε έναν κανονισμό που θα καλύπτει τις όλα τα κρατημέλη και τις ειδικέ ανάγκες τους. Αυτό που θέλω να πω βασικά είναι ότι έχουμε κάνει ως Κομισιόν και με αυτόν τον κανονισμό είναι να βοηθήσουμε και να ενισχύσουμε την περιφερειακή συνεργασία. Για, για σας δώσω ένα παράδειγμα, όχι από τον τομέα του αερίου, αλλά από τον τομέα του ηλεκτρισμού. Έχουμε συνεργαστεί πολύ στενά με το Ευρωπαϊκό Συντονιστικό Όργανα για να εξασφαλίσουμε ότι η κατάσταση η νησιωτική, ας το πούμε σε εισαγωγικά, που επικρατεί στην Ισπανία, που αφορά την Ισπανία, δεν θα επαναληφθεί στην περίπτωση του φυσικού αερίου. Ε, θα συνεργαστούν και τα κράτη-μέλη, όπως είπα, με, την ενίσχυση της Κομισιόν για, την περιφερειακή συνεργασία, να ενισχυθεί η περιφερειακή. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Είμαι πολύ σύντομος. Συμφωνώ με την ανάγκη για ένα νέο κανονισμό για ένα τόσο σοβαρό πρόβλημα. Και περνάω στο ερώτημά μου. Με ενδιαφέρει ιδιαίτερα το θέμα της συνεργασίας και της αλληλεγγύης. Τι μέτρα και τι αποδοτικά μέτρα προβλέπεται να ληφθούν προκειμένου να επιτευχθεί αυτός ο διπλός στόχος που κατά τη γνώμη έχει προτεραιότητα για να αντιμετωπιστεί μια σοβαρή κρίση. Απαιτεί μια Ευρώπη πιο ενωμένη και πιο ισχυρή. Απάντηση. Ο κύριος ε, ξανά. Εάν σας κατάλαβα καλά, πρέπει οπωσδήποτε να εξασφαλίσουμε την αλληλεγγύη μεταξύ μας αλλά και την, να είμαστε ε, να είμαστε υπεύθυνοι να εξασφαλίσουμε και την αλληλεγγύη και την ανάληψη των ευθυνών μας αυτό χρειάζεται, είναι προϋποθέσεις για τον κανονισμό κάθε εταιρεία κάθε κράτος μέλος θα πρέπει να αναλάβει τις ευθύνες του και να συμμετάσχει σε ένα σύστημα αλληλεγγύης. Και η αλληλεγγύη μπορεί να είναι ευρωπαϊκή, ευρωπαϊκή ένωση αλληλεγγύη, αλλά μπορεί να είναι και περιφερειακή αλληλεγγύη. Και απαντώ εν μέρη και στην προηγούμενη ερώτηση δεν έχει νόημα να μην υπάρχει αλληλεγγύη στην Ευρωπαϊκή Ένωση και όλοι οι μηχανισμοί ακριβώς αυτό προσβλέπουν στην ανάπτυξη και ενίσχυση της, του περιφερειακού στοιχείου, της περιφερειακής συνεργασίας. Ευχαριστώ ε, θερμά. Έχω μερικές ίσονος σημασίες ερωτήσεις. Θα ήθελα όμως να μου τις απαντήσετε. Πρόσεξα, κύριε Ρέτε, ότι σε αυτήν την έκθεση επιπτώσεων δεν αναφέρεται σχεδόν καθόλου ο ρόλος των επιχειρήσεων, του επιχειρησιακού τομέα στην, ε, ε, στο ξεπέρασμα της κρίσης. Ε, ότι προηγουμένως είχαμε συζητήσει και τον σημαντικό ρόλο, τη σημαντική συμβολή των επιχειρήσεων στο ξεπέρασμα, διότι βάσει αυτού μπορούμε και να προγραμματίσουμε από ποιον και με ποιον θα συνεργαστούμε για τις λύσεις. Επίσης, μέσα σε αυτή τη διαδικασία εφαρμόστηκαν οι κανόνες του έτους 2004, ο κανονισμός του 2004. βάσει του κανονισμού λοιπόν αυτού από το 2004 που διαπιστώσατε προβλήματα ε, ε, ε, εφαρμόστηκαν σωστά όλες οι διατάξεις όλες οι οι υποχρέωσεις, πού είναι τα κενά, πού παρουσιάστηκαν τα προβλήματα, πού κόλλησαν τα θέματα, γιατί πρέπει να εντοπίσουμε ακριβώς αυτά ε, τα προβλήματα ε, δεδομένου ότι προχωρούμε τώρα στον ε, νέο κανονισμό. Τι επιπτώσεις θα δημιουργηθούν εάν ο αγωγός Ναμπούκο, ο αγωγός της Βόρειας Θάλασσας μας προσφερθούν άλλη εναλλακτική αγωγή, άλλες εναλλακτικές λύσεις. Θα συνεχίσει να ισχύει το πρόβλημα που υπάρχει τώρα ή όχι. Άλλο θέμα. Είπατε επίσης ότι υπάρχει αυτή η εθελούσια, η εθελοντική συμβολή του, του βιομηχανικού τομέα. Ε, και βλέπω εδώ τη λέξη ανίκανη, untauglich στα γερμανικά, ανίκανη. Δεν βλέπω όμως καμία δικαιολόγηση του στοιχείου γιατί απεδείχθη ανίκανη. Και το τελευταίο τελευταία ερώτηση είναι ο καθορισμός του κόστους που σε ποια σημεία της αντίστροφης ροής ε, θα καθορίσουμε το κόστος διότι αναφέρεται εδώ το κόστος των επενδύσεων, πόσα θα είναι το κόστος των επενδύσεων για την εξασφάλιση της ροής στα κράτη-μέλη. Πού ακριβώς, σε ποια σημεία των έργων θα καθορίσουμε ε, το κόστος ε, στο κράτος μέλος Α ε, όπου ξεκινάει η αντίστροφη ροή στο κράτος μέλος Β τον αποδέκτη της αντίστροφης ροής σε ποια σημεία μάλιστα λέει ο Ρουτ Ε, ε, λέτε ότι είναι ίσονος σημασία. Εγώ θα έλεγα ότι είναι πολύ κέρυες οι ερωτήσεις αυτές. Το, τα προβλήματα κρύβονται στις λεπτομέρειες. Καταρχάς ο ρόλος των επιχειρήσεων. Ο, οι επιχειρήσει στην κρίση αυτή του, του φυσικού αερίου από τη Ρωσία στην αρχή του έτου, ήταν πάρα πολύ θετική η στάση των επιχειρήσεων. Το τονίσαμε αυτό πολλές φορές. Όμως οι εταιρείε είναι ιδιωτικοί φορείς και πολλές φορές ε, συναντούν εμπόδια απροσπέραστα και ομολογώ ότι στις συζητήσεις που είχαμε ήταν συγκλονιστικό να διαπιστώσουμε ότι δεν υπήρχε ούτε ίχνος ε, ε, προγράμματος αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών. Πολλά κράτη δεν είχαν καμία πρόβλεψη αντιμετώπισης τάκτων αναγκών. Επίσης, ορισμένα κράτη-μέλη αντιμετώπισαν την κρίση ε, σαν να βρίσκονταν ε, σαν να, προσπαθούσαν να φυλάξουν τις αποθήκες του φυσικού του αερίου πάνω στις οποίες καθόντουσαν και δεν ήθελαν να κουνήσουν. Δηλαδή, περίπου η στάση τους ήταν εμείς έχουμε το φυσικό αέριο, καθόμαστε πάνω του ακούνητη και δεν, δεν θέλουμε να αποχωριστούμε ούτε ένα ε, ποσοστό, ούτε, ούτε ένα ελάχιστο ποσοστό. Ε, ήταν λοιπόν και αυτή μια αντιμετώπιση ορισμένων κρατών μελών να μην συνεργαστούν. Ε, η, η απάντησή μου λοιπόν η μονολεκτική στο τι κάνουν οι εταιρείε για μένα είναι εσωτερική αγορά ενιαία αγορά. Την απάντηση της δίνει η εσωτερική αγορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τώρα, η οδηγία, οι κανόνες του 2004 δεν φτάνουν. Δεν φτάνουν και αυτό μπορούμε να το αποδείξουμε. Ε, το τεκμηριώνουμε, εάν κοιτάξετε πόσο διαφορετικά εφαρμόστηκαν τα διάφορα πρότυπα στα κράτη-μέλη, θα διαπιστώσετε ότι δεν φτάνουν. Ε, το αναφέρουμε αυτό στην έκθεση υποστήριξης ε, του κανονισμού για τους κανόνες του 2004. Βέβαια, επιδιώκουμε την διαφοροποίηση ε, και η των, των αγωγών. Ο αγωγός Βορείου Θαλάσσης, ο Βαλτική. Βαλτικής, ο αγωγός Ναμπούκο. Ε, εάν δούμε όλο το θέμα αυτό υπό την οπτική γωνία του νημείων 1, θα έχουμε διαφοροποίηση των, του εφοδιασμού. Αυτό όμως δεν αλλάζει την πραγματικότητα ότι μπορεί να δημιουργηθούν κρίσεις και ότι η Ευρώπη πρέπει να αντιδράσει. Πρέπει να έχουμε τη δυνατότητα αντιδράσεων. Τώρα, η ε, με, προαιρετικά μέτρα πρώτα να κοιτάξουμε τι μπορούν να κάνουν οι εταιρείες και εν συνεχεία στο, την, το επόμενο επίπεδο, τι μπορεί να κάνουν οι φορείς, το δημόσιο κλπ. Τα κράτη-μέλη. Ε, δεν μπορεί κανένας μόνος να αντιμετωπίσει τέτοιου είδου κρίσεις. Και ως υποσημείωση θέλω να πω ότι πριν από μερικού μήνες συζητήσαμε το θέμα των αποθεμάτων, πετρελαϊκών αποθεμάτων όπου έχουμε μία εντελώς άλλη φιλοσοφία σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση όπου υπό το πλαίσιο της ασφάλειας έχουμε προβλέψει αποθεματικά πετρελαίου. Και δεν έχουμε συμπεριλάβει ε, αυτές, ε, αυτά τα αποθέματα φυσικού αερίου στην ε, έκθεση αξιολόγησης επιπτώσεων, διότι πιστεύουμε ότι η αγορά και όλες αυτές οι ροές του φυσικού αερίου είναι τελείως διαφορετικές από το πετρέλαιο και το, την ασφάλεια εφοδιασμού. Η, αντίρροπος, ε, η αντίστροφη ροή ε, δείχνει ότι δεν πρέπει να εννοούμε πάντοτε μία μονοκατευθυντήρια ροή του φυσικού αερίου, αλλά πρέπει να ε, λάβουμε υπόψη και μια αντίστροφη ροή, έτσι ώστε το κόστος να ε, ε, πέφτει βεβαίως στις πλάτες του ωφελούμενου, του αποδοχέα. Αυτός ο οποίος χρησιμοποιεί την αντίστροφη ροή, ο αποδέκτης και ο χρήστης πρέπει να πληρώνει σε γενικό ευρωπαϊκό επίπεδο τώρα προσπαθώ να βρω ένα παράδειγμα η Γερμανία εδώ ενδεχομένως ο Γερμανός καταναλωτής ας πούμε δέχεται πληρών για την αντίστροφη ροή από την Πολωνία αλλά ο Ολλανδός ενδεχομένως που παίρνει την αντίστροφη ροή από τη Μεγάλη Βρετανία πληρώνει την αντίστοιχη προς τη Γερμανία. Πρέπει λοιπόν να το σκεφτούμε αυτό. Ε, και μία πάρα πολύ μικρή ερωτησούλα. Είπατε κύριε Ρίτε ότι υπήρξαν κράτη-μέλη. Αυτό μας ενδιαφέρει για την αξιολόγηση. Που που καθίσαν πάνω στα, στο φυσικό αέριο που έχουν και δεν δώσανε, δεν κονίσαν ρούπι. Ένα κράτος ήταν <laughs> αυτό που υπονοείται ή δύο. Επισήμως και δημοσίως δεν θέλω να εκφραστώ, λέει ο κύριος Ρούτε. Ευχαριστώ, λέει ο πρόεδρος, διότι το ερώτημα αυτό είναι σημαντικό, διότι πολλές φορές λαμβάνουμε πολιτικά, πρέπει να αναγκαστούμε να λάβουμε πολιτικά μέτρα, ενώ τα, τα προβλήματα είναι μικρά. Ο κύριος Βόμποντα επειδή είπε ο κ. Ρούτε ότι τα αποθέματα του φυσικού αερίου είναι διαφορετική ιστορία από τα πετρελαϊκά αποθέματα. Ναι, όμω βοηθούν, βοηθάει η ύπαρξη αποθεμάτων στο φυσικό αέριο. Μα το έδειξε η κρίση, έτσι δεν είναι. Ε, ωραία, δίνω τώρα πάλι το λόγο στην Κομισιόν για την ε, παρουσίαση του, του κανονισμού καθεαυτού. Okay, thank you very much. Uh, Ας έρθουμε στο σχέδιο κανονισμού. Θα σας επαναλάβω τις βασικές αρχές. Πρώτον, η πρόταση διασφαλίζει ότι η αγορά θα πρέπει να αντιμετωπίσει οποιαδήποτε διακοπή παροχής όσο και αν κρατήσει αυτό, διότι είδαμε ότι η εσωτερική αγορά είναι η πιο καλή εγγύηση για ασφαλή εφοδιασμό. οι εταιρείε να κάνουν τη δουλειά και να διασφαλίσουν τον εφοδιασμό. Βέβαια, η εσωτερική αγορά θα λειτουργήσει μόνο αν υπάρχει υποδομή, διαφάνεια της αγοράς και προληπτική διαχείριση της ζήτησης. Και έχουμε δει ότι υπάρχει έλλειψη στις υποδομές που εμποδίζει την εσωτερική αγορά να λειτουργεί σωστά. Έχουμε προβλήματα και με τη διαφάνεια Άρα θα πρέπει να δούμε πώς μπορεί να βοηθήσει η καλύτερη διαχείριση κρίσης. Επίσης, χρειάζονται κοινέ προδιαγραφές. Αν θέλουμε να έχουμε τους ίδιους κανόνες παιχνιδιού για όλους, θα πρέπει όλοι και η βιομηχανία, όλες οι εταιρείες παρατώσει, να ξέρουν ποιοι είναι οι κανόνες του παιχνιδιού. Οι κοινέ προδιαγραφέ λοιπόν είναι κομμάτι αυτών των κανόνων του παιχνιδιού. Εδώ έχουμε δύο προδιαγραφέ: Μία για τις υποδομέ νήμιον 1, και μία για τον εφοδιασμό αερίου για προστατευόμενους πελάτες. Φυσικά πρέπει να γίνει και ανάλυση κινδύνου σε κάθε επίπεδο, εθνικό, περιφερειακό ή της Ένωσης αφού θα εντοπιστούν οι κίνδυνοι υπάρχει ευελιξία που απαιτείται, επικουρικότητα δηλαδή για να αντιμετωπιστούν αυτοί οι κίνδυνοι μέσω της ζήτησης, μέσω περιφερειακής συνεργασίας κλπ. Με δύο λόγια δηλαδή στην πράξη τι απαιτείται. Πρώτον, αξιολόγηση του κινδύνου με βάση τις κοινέ προδιαγραφές για τις υποδομές νημιών 1 και για τον εφοδιασμό για τους προστατευόμενους πελάτες. Εφτά μέρες στην εποχή της εχμής του χειμώνα και 60 μέρες όταν υπάρχει ζήτηση το χειμώνα. Βέβαια, η εφαρμογή αυτών των προδιαγραφών σε κάθε χώρα θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη την δημορφία της κάθε χώρας. Δεν είναι 7 μέρες εχμή ή χειμώνα. Στην Ισπανία το ίδιο με τη Λιθουανία. Και αυτό πρέπει να οδηγήσει σε μέτρα προληπτικά ως προς τους κινδύνους και μέτρα έκτακτης, προγράμματα έκτακτης ανάγκης με τρία επίπεδα έγκυρη προειδοποίηση, συνογερμός, έκτακτη ανάγκη. Τα δύο πρώτα σημαίνει ότι η εσωτερική αγορά λειτουργεί, έκτακτη ανάγκη σημαίνει ότι οι εθνικές αρχές παίρνουν μέτρα ακόμα και κόντρα στην ενιαία αγορά. Πάντως αυτή η δουλειά δεν πρέπει να γίνεται μόνο σε εθνικό επίπεδο αλλά και σε περιφερειακό σε, και σε επίπεδο ένωσης αν απαιτείται. Όλος ο κανονισμός λοιπόν στηρίζεται πάνω σε αυτά. Νομική βάση άρθρο 95 Πλαίσιο εσωτερικής αγοράς γιατί σας είπα θέλουμε η εσωτερική αγορά είναι η πιο καλή εγγύηση για τον εφοδιασμό όσο πιο πολύ γίνεται χρονικά και δυνατόν για πάντα χωρίς να χρειάζεται να προσφύγουμε σε κρατικά μέτρα που θα πάνε κόντρα στην εσωτερική αγορά. Προληπτική δράση και μέτρα έκτακτης ανάγκης. Όλοι οι εμπλεκόμενοι πρέπει να λειτουργήσουν σε αυτό το πλαίσιο. Γι' αυτό χρειάζεται συνεργασία όλων και ενώ δημόσια αρχή, επιχειρήσεις αερίου, πελάτες στη χρήση αερίου ή αυτοί που παράγουν ηλεκτρισμό με αέριο, όλοι στο να καθοριστούν αυτά τα προγράμματα. Αυτή η διαδικασία πρέπει να κατευθύνεται από μία αρχή σε κάθε χώρα. Κάποιος πρέπει να κάθεται στο τιμόνι για αξιολόγηση κινδύνου για τα προληπτικά προγράμματα ή για τα προγράμματα έκτακτης ανάγκης. Έτσι δημιουργείται και αίσθημα ευθύνης που είναι βάση για την αγγελεγγύη. Ο καθένας θα αναλάβει έτσι τις ευθύνες του προκειμένου να οριστούν λύσεις από κοινού. Το εθνικό επίπεδο δεν επαρκεί, χρειάζεται και περιφερειακή συνεργασία. Και η Κομισιόν θα βοηθήσει στη διαδικασία αυτή. Να υπάρχει αυτή η περιφερειακή διάσταση. και έτσι δημιουργείται ένας δυναμισμός που θα ενισχύσει τη συνεργασία και την αλληλεγγύη. Πρέπει να υπάρχει σαφήνεια στο περιεχόμενο και στο πώς θα ε, ξεκινήσει η εφαρμογή των προγραμμάτων έκτακτης ανάγκης. Θα πρέπει να αναφερούνται τα προγράμματα από την Κομισιόν σε διαβούλευση φυσικά με την ομάδα συντονισμού για το αέριο και με τους άλλους φορείς. Επίσης προτείνουμε να ενισχυθεί η ομάδα για τον συντονισμό του αερίου Gas Coordination Group όπου θα έχουμε και εκπροσώπους των κυβερνήσεων και εκπροσώπους της βιομηχανίας. Δείκτης νήμιον 1. Θα τον εξηγήσουμε λίγο. Καταρχήν είναι μια αρχή που είναι γνωστή από τον κλάδο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. Είναι ο βασικός κανόνας εκεί. Ισχύει όμως και από μερικές χώρες όπως η Ισπανία και για το αέριο. Σημαίνει αν η πιο μεγάλη υποδομή αποτύχει η υπόλοιπη υποδομή να παρέχει επαρκή εφοδιασμό για να καλύψει τον εφοδιασμό με αέριο. Δηλαδή είναι ένας δείκτης στον οποίο πρέπει να μπουν νούμερα και στοιχεία σε σχέση με το δυναμικό του συστήματος αερίου. Φυσικά, η κάθε χώρα έχει διαφορετική υποδομή. Μερικές χώρες έχουν ιστορική παραγωγή ή μεγάλη ικανότητα αποθήκευσης. Μπορεί να έχουν πολλούς αγωγούς που να τροφοδοτούν την αγορά από διάφορες κατευθύνσεις. Με πολλούς δηλαδή ε, από εφοδιασμό από πολλές προελεύσεις. Άλλοι είναι πιο περιορισμένοι και στην υποδομή, άρα είναι πιο εκτεθειμένοι σε κινδύνους. Το είδαμε αυτό στην πράξη. Εν πάση περιπτώσει όμως, είναι κοινή αναφορά για όλους. Και λαμβάνεται υπόψη έτσι η κατάσταση κάθε χώρας για να μπορούμε να συγκρίνουμε την ασφάλεια σε κάθε χώρα. Και εδώ έχουμε ένα στοιχείο ευθύνης που είναι βάση για αλληλεγγύη. Μπορεί να υπολογιστεί αυτός ο δείκτης σε εθνικό επίπεδο, σε περιφερειακό επίπεδο ή σε επίπεδο ένωσης. πάτε όποιο μέγεθος θέλετε και αξιολογήστε αν μπορείτε να ε, μετριάσετε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τους κινδύνους που εντοπίσατε στην αξιολόγηση κινδύνων. Φυσικά προσφέρουμε και τη δυνατότητα στα κράτη-μέλη και ενώ όλους τους φορείς του αερίου σε κάθε χώρα να ορίσουν τη σωστή λύση. Μπορεί να αυξηθεί ας πούμε το αποθηκευτικό δυναμικό με διάφορα τερματικά επιπλέον παραγωγή για αυτούς που παράγουν αντίστροφη ροή και διαχείριση της ζήτησης με αλλαγή χρήσης φερρυπίν του καυσίμου Κάναμε μια προσωμείωση του Δίκτυν Νιον 1 που στηρίζεται σε στοιχεία που πήραμε ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια της κρίσης και μετά και από μια εταιρεία IHS. Γιατί και εμείς δεν έχουμε επαρκή στοιχεία. Γι' αυτό σας μίλησα πριν για έλλειψη διαφάνειας. Με βάση τα στοιχεία που έχουμε κάνουμε μία προσωμείωση των ήμιων ένα για κάθε χώρα. Είναι ενδιαφέρον να αρχίσουμε από το άκρα δεξιά που βλέπετε αν το εφαρμόσετε σε επίπεδο ένωσης η ένωση είναι μάλλον ασφαλής όσον αφορά τον εφοδιασμό. Υπάρχουν πολλά σημεία εισόδου, διαφοροποίηση δηλαδή στον εφοδιασμό, αλλά να περάσετε σε κάθε χώρα μέλος βλέπετε ότι μερικές διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο από ό,τι άλλες. Πήραμε τα στοιχεία όσοι έχουν σήμερα. Αυτό είναι το μπλε στο διάγραμμα. Και κάνουμε μία προσωμείωση ποια θα ήταν η κατάσταση αν τα προγράμματα που είναι τα προγράμματα ανάκτησης που εγκρίθηκαν από το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο πρόσφατα τι θα μας έδιναν ως αποτέλεσμα προγράμματα σύνδεσης ή αντίστροφων ροών. Εδώ βλέπετε ότι η κατάσταση βελτιώνεται για κάποιες χώρες, όχι για όλες. Αυτός ο δείκτης νήμιον 1 δεν είναι ένα μηχανικό σύστημα. Το πιο καλό παράδειγμα είναι η Φιλανδία. Στη Φιλανδία έχουμε μια χώρα που έχει ένα μόνο από τη Ρωσία κόβει το γόγος, σταματάει το αέριο. Αλλά στη Φιλανδία το ξέρουν αυτό και υποχρέωσαν όλους τους καταναλωτές αερίου να αλλάξουν καύσιμο. Στη ρήψη που δεν έχουν αέριο μπορούν να αντικαταστήσουν με άλλο καύσιμο. Αυτό είναι βέβαια εξαίρεση. Αλλά μας δείχνει ότι πώς μπορεί να ληφθεί υπόψη το στοιχείο επικουρικότητα. Κοινωτική διάσταση. Μερικοί ρώτησαν τι κάνει η κοινότητα. Είδαμε ότι μία διακοπή μπορεί να οδηγήσει σε κοινωτικό πρόβλημα. Η κοινότητα πρέπει να αντιδράσει δηλαδή συντονισμένα. στην περίπτωση αυτή η Κομισιόν θα πρέπει να φροντίσει τα προγράμματα που υπάρχουν, τα προληπτικά και έκτακτης ανάγκης, να λάβουν υπόψη την διάσταση της γειτονικέ χώρες κλπ. Αυτός είναι ο ρόλος της Κομισιόν για περιφερειακά προγράμματα. Στη διαδικασία αυτή η κοινότητα φυσικά θα έχει διαβουλεύσεις με την ομάδα συντονισμού και υπάρχει και ένα μέτρο που είναι λίγο πιο δύσκολο αλλά εξίσου σημαντικό. Σε έκτακτες περιπτώσεις η Κομισιόν μπορεί να ζητήσει από τα κράτη-μέλη να μην πάρουν αρνητικά μέτρα, αρνητικά για γειτονικέ χώρες. Καλό θα είναι να αποφεύγονται τέτοια είδους μονόπλευρα μέτρα που δημιουργούν ζημιά σε γειτονική χώρα και η αύξηση της διαφάνειας απαιτείται. Αντίστροφες ροές. Συζητήθηκε αυτό αρκετά. Αντίστροφη ροή δίνει περισσότερη ευελιξία στο σύστημα μεταφοράς αερίου Οι ανατολικές χώρες καλύπτονται από αγωγούς που κινούνται από την Ανατολή προς τη Δύση και δεν μπορούν να πάνε από τη Δύση προς την Ανατολή. Όταν είναι λοιπόν άδειοι γιατί δεν έχετε τίποτα από την Ανατολή, δεν μπορούν να λειτουργήσουν με αέριο που έρχεται από τη Δύση. Το είδαμε αυτό. Και είδαμε ότι μέσα σε δύο εβδομάδες οι Τσέχοι και οι Σλοβάκοι κατάφεραν να αντιστρέψουν τη ροή. Που σημαίνει, δεν το δεν ξέραμε ότι μπορεί να συμβεί αυτό πριν, αυτό έδειξε δημιουργικό πνεύμα των μηχανικών. Μέσα σε δύο εβδομάδες αντέστρεψαν τη ροή. Χρήσιμο για τη Σλοβακία. Η Βουλγαρία και η Ελλάδα επίσης προς το τέλος της κρίσης κατάφεραν και αυτοί να μεταφέρουν αέριο από την Ελλάδα προς τη Βουλγαρία. Δεν μιλάμε για τεράστιες επενδύσεις. Είναι κάτι που πρέπει να μελετηθεί και υπάρχει μια μελέτη στη διάθεσή σας αν θέλετε όπου έχουν εντοπίσει στη μελέτη αυτή 43 ειδικά προγράμματα για αύξηση της ασφάλειας εφοδιασμού. Μικρές επενδύσεις 1 έως 5 εκατομμύρια φτηνά αν το συγκρίνουμε με το πώς θα στοιχήσουν νέοι αγωγοί, όπου μιλάμε για εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ. Πιστεύουμε λοιπόν τα προγράμματα αντίστροφη ροή είναι σημαντικά και πρέπει να τους βοηθήσουμε και με κοινωνικά κονδύλια. Και φυσικά πρέπει να υπάρχουν και κριτήρια κόστους απόδοσης και η υποχρέωση όλα αυτά να εφαρμόζονται με προσοχή. Τα ωφέλη αντίστροφων ροών. Για να τελειώσουμε, για να δούμε ποια χώρα ε, από τις αλλαγές αυτές. Βλέπετε ε, τα βέλη ξεκάθαρα. Αν μπορέσουν να λειτουργήσουν από την κατεύθυνση από δυσμάς προς Ανατολάς θα βοηθηθούν πολύ ε, αυτές οι χώρες, οι περισσότερες, από τις οποίες επλήγησαν ε, αρκετά ε, τον Ιανουάριο. Το ίδιο ισχύει για την Νότιο-Ανατολική Ευρώπη. Αν έχουμε διπλής κατεύθυνσης ε, αγωγούς και ροές μεταξύ Ελλάδας, Βουλγαρίας και Ρουμανίας, θα επιτραπεί πολύ καλύτερα η αντιμετώπιση κοπής παροχής φυσικού αερίου και ροής από την Ουκρανία, για παράδειγμα. Έχουμε και άλλο παράδειγμα για την Ελλάδα και τη Βαλκανική. Ε, δηλαδή για να σας δείξω ότι η κρίση του Δεκεμβρίου οδήγησε τον κλάδο να αναζητήσει λύσεις και να αναρωτηθούμε. Μπορούμε πολύ γρήγορα να κάνουμε κάτι. Εάν ξαναζήσουμε τέτοια κρίση τους ερχόμενους μήνες, ναι. Έχει γίνει πολλή δουλειά όντως και βγάλαμε τα συμπεράσματα και τα διδάγματά μας και προσπαθεί και ο κλάδος στο μέλλον να μετριάσει όσο γίνεται και να ακουφίσει από ενδεχόμενη κρίση. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ. Εκτενέστατη για αυτή η παρουσίαση. Θα ήθελα να δώσω πρώτο το λόγο στον εισηγητή μας, τον κύριο Βινταλ Κουαδράς. Παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Είχα κάποιες πρώτες ανταλλαγές απόψε με μέλη τη Επιτροπής μα για την νομοθετική αυτή πρόταση και έχω την ικανοποίηση να σας ε, λέγω ότι η αντίδραση των μελών τη Επιτροπής μας ήταν θετική σε σχέση με την πρόταση Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Όντως η Κομισιόν μας κάνει μια καλή πρόταση και θα προσπαθήσουμε, όπως πάντα κάνουμε, να βελτιώσουμε. Αλλά σε γενικές γραμμές ανταποκρίνεται και απαντά όχι μόνο στις ανησυχίες και τα μελήματα του Κοινοβουλίου στο παρελθόν, αλλά και στην πραγματικότητα του προβλήματος. Αν καταφέρουμε να φέρουμε αυτόν τον κανονισμό σε αίσιο πέρας και να εφαρμοστεί όμως ε, σε εύλογο χρόνο, ε, τότε η Ευρωπαϊκή Ένωση θα μπορέσει να μειώσει σημαντικά τη ευάλωτη θέση της ε, απέναντι σε ενδεχόμενες διαταραχές στη βαροχή αερίου και διακοπές στο μέλλον. Υπάρχουν συγκεκριμένα μέτρα τα οποία ορίζουμε υποχρέωση να έχουμε προγράμματα αντιμετώπισης κρίσεων και εκτάκτων αναγκών σε τοπικό επίπεδο, περιφερειακό, εθνικό και ευρωπαϊκό, έγκαιρη προειδοποίηση σε διάφορα επίπεδα, σαφής ορισμός ε, των υποχρεώσεων που έχει κάθε κλάδος, βελτίωση της ε, διαφάνειας, μέθοδος νη 1, για να διατηρηθεί η παροχή σε περίπτωση που διακοπεί από τη βασική πηγή. Εν πάση περιπτώσει, όλα αυτά τα στοιχεία που μας ε, λέτε μας φαίνονται εύστοχα. Τώρα, υπάρχουν κάποιοι τομείς ε, όμως που θεωρούμε ότι χωράει βελτίωση η πρόταση. Για παράδειγμα, μια ανησυχία που έχουμε εμείς είναι ότι δεν ορίζεται σαφώς πότε τα κράτη-μέλη θα μπορέσουν να προχωρήσουν σε μηχανισμούς που δεν είναι της αγοράς. Λέγεται ότι όταν θεωρούνται αναπαρκή ε, τα μέσα της αγοράς για να αντιμετωπιστεί η κρίση. Αλλά όπως έχει ο κανονισμός αυτή τη στιγμή, δεν μπορεί κανείς να αποκλείσει ε, ότι κάποια χώρα μέλος θα πάρει την απόφαση πριν εξαντλήσει όλες τις δυνατότητες της αγοράς. Έτσι. Δηλαδή, τι εννοώ. Βεβαίω και δεν αντιτιθέμεθα στο θέμα αυτό. Υπάρχουν ε, καταστάσεις που ε, απαιτούν ε, κρατική παρέμβαση, αλλά θα πρέπει να κλειδώσει έτσι το κείμενο ώστε να μην χωράει καμία αμφισημία. Ένα άλλο θέμα που με ανησυχεί και συνδέεται με αυτό είναι η υποκατάσταση του καυσίμου. Fuel shooting το λένε αυτό. Αλλαγή καυσίμου. Υπάρχουν συμβατικές υποχρεώσεις, μεν, από την άλλη όμως υπάρχει και το θέμα ε, εξαναγκασμού γιατί έχουμε επιπλέον εκπομπές ε, διοξιδίου του άνθρακα. Δεν μπορούμε να ζητήσουμε από τη βιομηχανία να επομιστεί ένα τέτοιο κόστος που θα αυξάνει τις εκπομπές αερίου και να επομίζονται ένα κόστος για το οποίο δεν φταίνε. Δηλαδή, θα πρέπει να δούμε ποιο θα πληρώσει αυτά τα δικαιώματα εκπομπών, πώ θα σταθμίζονται και εδώ δεν χωράει καμία σύγχυση. Υπάρχουν κάποιες παράγραφοι του κανονισμού που αφορούν ανταλλαγή πληροφοριών. Πολύ σημαντικές αυτές ε, στην πρόταση. Μεν. Πλην όμως, ξέρετε ότι θα υπάρξουν πολλά κράτη-μέλη που θα έχουν μεγάλες επιφυλάξεις και αντιστάσεις. Το ίδιο ισχύει και με τις εμπορικές συμφωνίες. Εδώ θα πρέπει λίγο περισσότερο να χτενιστεί το κείμενο, να ξεκαθαριστεί. Να υπάρχει μια ρήτρα, ας πούμε, εμπιστευτικότητας. Για να ε, διασκεδαστούν οι αφιβολίες. Η ομάδα συντονισμού για το φυσικό αέριο νομίζουμε θα πρέπει να έχει ενισχυμένο ρόλο ε, σε σχέση και με τα εθνικά σχέδια εκτάκτου ανάγκης κυρίως επειδή, όπως είπατε κι εσείς, ε, αυτό έχει αποδειχθεί αποτελεσματικό στην πράξη σε προηγούμενες κρίσεις. Και επίση το όργανο αυτό, η ομάδα συντονισμού για το φυσικό αέριο, προσφέρεται για το περιφερειακό συντονισμό. Δηλαδή, μπορεί λοιπόν να συμπληρωθεί ο ρόλος ε, ο βασικός αυτός της Ευρωπαϊκής Επιτροπής από μια ενίσχυση της ομάδας συντονισμού για το αέριο. τι είναι οι προστατευόμενοι πελάτες. Και αυτό επίσης θα πρέπει να το συζητήσουμε ως ορισμό, διότι ανάλογα με την κατάσταση. Δηλαδή όσο διευρύνεται ο αριθμό των πελατών αυτών, η μέθοδος νη ε, πλην 1 εφαρμόζεται με μεγαλύτερη ή μικρότερη εμβέλεια. Και όπως είναι φυσικό αυτό έχει επιπτώσεις και για τις επενδύσεις και για το κόστος που είναι ενδεχομένως αρκετά υψηλές. Έτσι λοιπόν, έχουμε ενώπιό μας ένα κανονισμό που προσπαθεί να μας ε, βγάλει από ακραίες καταστάσεις με οικονομικές, πολιτικές και ανθρωπιστικές συνέπειες εξαιρετική σημασίας. Ας μην ξεχάσουμε και αυτή την τελευταία διάσταση. Στην τελευταία κρίση ε, προμήθειας είχαμε καταστάσεις ε, που από ανθρώπινης πλευράς ήταν δραματικές, ήταν τραγωδίες για κάποια κράτη-μέλη. Και δεν μπορούμε να το ξεχνάμε αυτό. Θα πρέπει να το έχουμε πάντα στο μυαλό μας όταν συζητούμε για τον κανονισμό αυτό. Καταρχήν λοιπόν κύριε Πρόεδρε έχω την εντύπωση ότι η Επιτροπή μας υποστηρίζει την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να είναι κανονισμός δηλαδή και όχι οδηγία και η νομική βάση που χρησιμοποιείται θα πρέπει να είναι η συναπόφαση βεβαίως. Από τότε που τέθη ισχύ αυτή η ρύθμιση έχει κυλήσει πολύ νερό στα βλάκι, έχουν αλλάξει πολλά πράγματα και έχουμε όλη ευθύνη που μας υποχρεώνει να προχωρήσουμε ακόμα παραπέρα. Αυτό λοιπόν προσπαθεί να κάνει αυτός ο κανονισμός και εμείς όπως πάντα θα βάλουμε τα δυνατά μας και θα κάνουμε ό,τι μπορούμε. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ. Ο συνάδελφος κύριος Ριτζιπ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα ήθελα να πω ότι χαιρετίζω την ε, πρόταση της ε, Επιτροπής, της Κομισιόν, σε αυτό το σχέδιο κανονισμού για την ασφάλεια του εφοδιασμού φυσικού αερίου. Είναι ένα βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση. Αυτό το βήμα ίσως το εμπνεύστηκα η Κομισιόν μετά την κρίση του Ιανουαρίου. Εμείς στην Πολωνία είχαμε ε, δεν είχαμε τόσο μεγάλη ε, επίπτωση από την κρίση. Ε, ορισμένα μικρά προβλήματα κατά τη διάρκεια της κρίσης, αλλά τα προβλήματα άρχισαν όταν η κρίση τελείωσε, μετά τον Ιανουάριο. Επειδή Λόγω της κρίσης, ένας από τους προμηθευτές φυσικού αερίου έκλεισε και αυτός ο προμηθευτής ε, παρέσχε 15% του φυσικού αερίου της Πολωνίας και έπρεπε να βρούμε το φυσικό αέριο αυτό από αλλού γιατί σταμάτησε να λειτουργεί. Ε, ευτυχώς ξεπεράσαμε αυτή την κρίση και δεν έχουμε άλλα προβλήματα μετά τον Ιανουάριο. Το θετικό αποτέλεσμα της κρίσης ήταν το εξής. Μέσα σε δύο εβδομάδες οι προμηθευτές αερίου μπόρεσαν να παράσχουν το αναγκαίο φυσικό αέριο στην Τσεχία και τη Σλοβακία. Και θετικό ήταν επίσης η αλληλεγγύη την οποία δείξαμε στο να βοηθήσουμε ε, άλλες περιοχές που είχαν προβλήματα. Όμως υπήρχαν ελλείψεις και στις διαδικασίες και στην, στις υποδομές. Ελλείψεις που πρέπει να καλυφθούν, πρέπει να αντιμετωπιστούν. Γι' αυτό ακριβώς ε, χαιρετίζω την πρόταση της Κομισιόν. Επίσης, σχετικά με την ενεργειακή πολιτική, η ενεργειακή αλληλεγγύη είναι ένα στοιχείο το οποίο ζητούμε εδώ και χρόνια εμείς στην Πολωνία. Και γι' αυτό εγώ ως Πολωνός Ευρωβουλευτής είμαι πολύ ευτυχής που βλέπω αυτή την πρόταση στο τραπέζι μας. Θα ήθελα να θέσω τρεις ερωτήσεις που είναι απολύτως σχετικές με το θέμα. Η Κομισιόν το ανέφερε, ανέφερε αυτό που θέλω να ρωτήσω στο πρώτο μέρος της συζήτησης. Είναι αυτός ο δείκτης, αυτό το πρότυπο, νήμιον ένα. Ο κανονισμός ε, θέτει πρότυπα ε, για την υποδομή και λέει τρία χρόνια θα χρειαστούν, τρία χρόνια είναι η πληθυσμία για τις υποδομές που πρέπει να κατασκευαστούν και δύο χρόνια για τις υπάρχουσες υποδομές προσαρμογής δηλαδή του δείκτη σε αυτές τις υποδομές. Για, την υπάρχουσα, ε, ε, για τις υπάρχουσες υποδομές πιστεύω ότι τα δύο χρόνια είναι πολύ, είναι υπερβολικό χρονικό διάστημα ε, για τις υποδομές όμως που δεν υπάρχουν ακόμα και που πρέπει να δημιουργηθούν πιστεύω ότι τα τρία χρόνια δεν είναι επαρκή. Θα πρέπει ίσως να ρωτήσουμε τους κατασκευαστές, τους ενδιαφερόμενους του κλάδου αν φτάνουν τα τρία χρόνια. Εν συνεχεία, στο άρθρο 10 αναφέρεται η κατάσταση, έκτακτη κατάσταση κινδύνου και αναφέρει την, ε, ε, ότι ο καθεστώς έκτακτης ε, ανάγκης μπορεί να δηλωθεί όταν δεν υπάρχουν, ε, διακοπούν οι προμήθειες ε, σε, ένα κράτος μέλος ή όταν οι προμήθειες σε φυσικό αέριο είναι ανεπαρκείς. Ε, αυτή λοιπόν η κατάσταση έκτακτης ανάγκης, εάν παρουσιαστεί σε ένα κράτος και εάν εφαρμόσουμε κατά λέξη τον κανονισμό, δεν θα μπορέσει να παρεσχεθεί η βοήθεια από άλλες χώρες πώς θα εξασφαλίσει την παροχή βοήθειας από τις άλλες χώρες σε περίπτωση τέτοιας έκτακτης ανάγκης την οποία καλεί ένα μόνο κράτος μέλος. Ε, μία άλλη μου παρατήρηση αφορά τις πληροφορίες τις οποίες οι ε, διαφερόμενοι πρέπει να δηλώσουν. Εφόσον θέλουμε να κάνουμε μία αξιολόγηση ποιες πληροφορίες θα μπορέσουμε εμείς να αξιολογήσουμε, ποιες θεωρούνται πιστευτικές, παραδείγματο χάρη ότι είναι εμπορικό ή βιομηχανικό, καλύπτονται από την βιομηχανική εμπιστευτικότητα ή ε, είναι έμπιστα στοιχεία αυτά στο εμπόριο και δεν μπορούν να δηλωθούν. Ο κύριος Σβόμποντα. Ευχαριστώ. Ως ε, σκιώδης εισηγητής θέλω να κάνω μερικές γενικές παρατηρήσεις. Αυτό το κανονισμό, το σχέδιο κανονισμού πρέπει να το μελετήσουμε μαζί με άλλα στοιχεία ενεργειακής επάρκειας, εφοδιασμού, διαφοροποίηση, Ουκρανία, αυτά τα οποία έχουμε αλλάξει, αυτά τα οποία θέλουμε να εφαρμόσουμε για να καταλήξουμε σε ένα σωστό αποτέλεσμα Όσον αφορά τον ενεργειακό χάρτη, μπορούμε να πούμε ότι δεν θα ε, ε, δεν θα επικυρωθεί αυτό και διότι έχουν δηλώσει πολλοί ότι δεν είναι πρόθυμοι να επικυρώσουν αλλά εν πάση περιπτώσει πρέπει να τα δούμε συγκεντρωτικά μας σε συνδυασμό και με άλλους κανονισμούς εάν λοιπόν περάσει ένας τέτοιος κανονισμός τα προβλήματα της ασφάλειας του εφοδιασμού θα μπορούν, ε, ο κανονισμός αυτός μπορεί να ενεργήσει ως μοχλός πίεσης κατά ενός κράτους, διότι οπωσδήποτε δεν θα του αρέσει ενός κράτους μέλος να υποστεί μια τέτοια εκβιαστική πίεση σε περίπτωση που θέλει να αλλάξει την ε, ροή. Επίσης, ε, ο ρόλος του ιδιωτικού τομέα εδώ πρέπει να διευκρινίσουμε ο Πρόεδρος, εγώ και άλλα μέλη που έχουμε χειριστεί την οδηγία του αερίου, πάντοτε λέγαμε ότι το αέριο δεν είναι το ίδιο, ίδιο και αυτό με το πετρέλαιο, άλλο το άλλο το άλλο. Όμως πρέπει και εδώ να συζητήσουμε με τους ε, ιδιωτικού φορείς που έχουν διαπιστώσει ότι υπάρχουν δυσκολίες ε, και γι' αυτό το λόγο πρέπει να διευρύνουμε τις επαφές μας. Πρέπει να, ε, να είναι δημόσιες οι πηγές πληροφόρησης. Εδώ υπάρχει έντονη αντίδραση. Η Κομισιόν πρέπει να έχει μια γενική επισκόπηση των επαφών, ποιος και που, και από πού, για να μην, και να μην αντιμετωπίζει μια γενική άρνηση πολλοί έρχονται και μας λένε το ένα και το άλλο, αλλά ουσιαστικά ε, για το χαρακτήρα του κανονισμού είναι σημαντικό και ο συγητής το αναγνωρίζει αυτό, είναι έμπειρος, το κοινοβούλιο να λειτουργήσει γρήγορα, ταχύτατα, διότι πιέζει ο χρόνος, ο πρόεδρος. Ευχαριστώ και Ζώγοτο. Ο κύριος Έντσου. Ευχαριστώ. Αγαπητοί συνάδελφοι, το σχέδιο κανονισμού το οποίο συζητούμε σήμερα προβλέπει ε, πολλές διατάξεις για να αντιμετωπιστεί μία κρίση. Θα πρέπει όμως οι υπηρεσίες ε, για ε, την ε, χρησιμοποίηση των πρωτοπαραγωγικών πηγών θα πρέπει να λειτουργούν καλύτερα αλλά και υπάρχει και η Ένωση Προμηθευτών Φυσικού Αερίου και με αυτήν πρέπει να έρθουμε σε επαφή. Άρα λοιπόν σωστά η ότι πρέπει να διευρύνουμε το δίκτυο επαφών. Είναι σωστό ότι ορισμένες διατάξεις του κειμένου θα πρέπει να ε, βελτιωθούν ε, όσον αφορά την ανταλλαγή πληροφοριών με την Κομισιόν ε, και την ομάδα συντονισμού φυσικού αερίου και τις αρμόδιες τοπικές αρχές, όπως προβλέπεται στο άρθρο 12 του κανονισμού. Ε, πιστεύω ότι η Κομισιόν θα πρέπει για να ληφθούν τα κατάλληλα μέτρα θα πρέπει να επιβάλλει μια απόλυτη διαφάνεια σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης και πρέπει να μιλήσουμε α, να διαθέτουμε αυτοματοποιημένα συστήματα ε, και να μπορέσουμε να ξεπεράσουμε γραφειοκρατικά προσκόμματα σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης πρέπει να μπορούμε να αντιδρούμε γρήγορα, τα ταχύτερον, διότι διαφορετικά και πιστώσεις θα χάνουν, και κονδύλια θα χάνονται και, ε, το, και της Ευρώπης θα υποφέρει. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Αυτός εδώ ο κανονισμός είναι ένα θετικό βήμα. θετικό βήμα, ιδιαίτερα σε σχέση με την κρίση του Ιανουαρίου. Αλλά πρέπει να έχουμε επίγνωση του γεγονότος ότι η κρίση αυτή μπορεί να επαναληφθεί και η Ευρώπη θα πρέπει να είναι έτοιμη Επειδή η υπόθεση αυτή είναι πολύ σημαντική, γιατί από αυτό εξαρτάται η παραγωγή ηλεκτρισμού, η θέρμανση, η πρώτη ύλη για τη βιομηχανία, το καύσιμο των μεταφορών. Πρέπει να έχουμε επίγνωση το ότι στις μεγάλες συμμαχίες του αερίου στηρίζεται η γεωπολιτική ισορροπία των κρατομελών για τις προσεχείς δεκαετίες. Παραδείγματο χάρη, τα τρία, οι τρεις ε, αεριοαγωγοί, Ναμπούκο, Nord Stream και South Stream, που προορίζονται να μεταφέρουν φυσικό αέριο προς πολλές χώρες της Ευρώπης, είναι ένα παράδειγμα μιας μάχης κατά κάποιο τρόπο που αφορά τη γεωπολιτική ισορροπία της Ένωσης και το βαθμό αυτονόμησής της ως προς τρίτες χώρες. Και γιατί τα λέω αυτά. Μεταξύ των ορυκτών καυσίμων, το φυσικό αέριο έχει την πιο μικρή εκπομπή διοξιδίου του άνθρακα. Άρα είναι αναπόσπαστο στοιχείο για τη μετάβαση προς μια οικονομία που να στηρίζεται σε πηγές ενέργειας καθαρές και ανανεώσιμες. Το ερώτημα λοιπόν και η ανησυχία αν θέλετε η δική μου και σας την παρουσιάζω είναι γενικού χαρακτήρα αναφέρεται στην ευρωπαϊκή διάσταση εφοδιασμού σε αέριο αν δεν γίνουν επενδύσεις μεγάλες για υποδομή για ασφάλεια για τον εφοδιασμό η Ευρώπη χωρίς αυτές τις επενδύσεις διατρέχει τον κίνδυνο να αυξηθεί η εξάρτησή της από μία χώρα, μία άλλη χώρα, στην περίπτωσή μας από τη Ρωσία. Αν το Ναμπούκο για την Ευρώπη ήταν μια μεγάλη ευκαιρία και η πρόσφατη συμφωνία Ιταλία-Τουρκία-Ρωσία υπάρχει κίνδυνος να υπονομεύσει το πρόγραμμα αυτό, αυτή την προοπτική. Ένα σημαντικό κομμάτι εφοδιασμού της Ευρώπης δηλαδή να εξακολουθήσει να εξαρτάται από μία χώρα. Αυτό είναι σχόλιο και ερώτημα. Και πρέπει να ξεκινήσει συζήτηση για το θέμα αυτό. Με πρωτοβουλίες που θα εμποδίσουν να επαναδιαγραφούν οι γεωπολιτικές ισορροπίες στην Ευρώπη. Συμπερασματικά, καλά είναι τα μέτρα του σχεδίου του κανονισμού που μας επιτρέπουν να κάνουμε ένα θετικό βήμα και αν υπάρχει νέα έκτακτη ανάγκη σε επίπεδο ένωσης αλλά πρέπει να προσέξουμε μην τυχόν η Ευρώπη εξαρτηθεί από μία μόνο χώρα για εφοδιασμό. Αδιαμφισβήτητα το θέμα της εμπιστοσύνης, της αγγελεγγύης, της συνεργασίας είναι πολύτιμο. Ευχαριστώ. Πρόεδρος, ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ο, ο κύριος Βαλτσίτης. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα να, να πω στην Κομισιόν και στους εκπροσώπους της ότι αυτό το κείμενο, αυτό το έγγραφο, είναι ισόρροπο και χαίρομαι που αναφέρει το πρόβλημα των λεγόμενων νήσων φυσικού αερίου διότι αυτό έχει άμεση επίπτωση στα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε ε, όσον αφορά την πολιτική εξάρτηση με μονομένο προμηθευτό φυσικού αερίου. Το, το μέγεθος προβλήματος της εξάρτησης. Ε, ο εφοδιασμός ε, σε φυσικό αέριο εξαρτάται και από τις τιμές των άλλων ε, ε, ε, φυσικών πόρων. Η τιμή του φυσικού αερίου εξαρτάται και από την τιμή του ηλεκτρικού. Αυτή τη στιγμή χτίζεται ένα τεράστιο εργοστάσιο παραγωγής στο Καλίνιγκραντ. Θα ήθελα λοιπόν να ρωτήσω ένα πυρηνικό εργοστάσιο στο Καλίνιγκραντ. Να αν η Κομισιόν μπόρεσε, θα μπορούσε να είχε προβλέψει την κρίση αυτή από τη Ρωσία και αν μπορεί να προβλέψει από ποια ενδεχόμενη πηγή παροχής φυσικού αερίου θα προκύψει η επόμενη κρίση για τα ευρωπαϊκά ε, κράτη. Ευχαριστώ. Ο Σύναφος Κάρινς. Ε, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να κάνω μια ερώτηση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για ε, τις λεγόμενες ενεργειακές νήσους, όπως είπε και ο συνάδελφος προηγουμένως. Η Λετωνία, σε ό,τι αφορά το φυσικό ε, αέριο και την προμήθεια και τον ανεφοδιασμό, είναι πάρα πολύ ασφαλής χώρα. Σχεδόν καμία επίπτωση δεν είχαμε από τα γεγονότα του Ιανουαρίου, ε, γιατί έχουμε αποθεματικό, αποθήκες υπόγειες για δύο χρόνια και από εκεί μπορούμε να τροφοδοτούμε και τα γειτονικά μας κράτη, τη Λιθουανία και την Εστονία, αλλά και την ίδια τη Ρωσία στην περιοχή γύρω από το, την Αγία Πετρούπολη. Πολλές φορές από τη Λετωνία παίρνει ε, φυσικό αέριο και έχουμε αντίστροφη ροή λοιπόν προς Ανατολάς. Θα μπορούσα να σας πω εδώ ότι ε, είμαστε σε πολύ καλή κατάσταση αφενός, αλλά αν καθίσουμε και σκεφτούμε και προβληματιστούμε, Πρέπει να σας πω ότι ολόκληρη η υποδομή του φυσικού αερίου για μας είναι ε, στα χέρια της Gazprom. Δηλαδή είτε ανήκει αποκλειστικά στη ε, Gazprom είτε έχει προνομιακά δικαιώματα για χρήση για κάποια χρόνια. Θα πρέπει αυτά να λυθούν. Καταλαβαίνω βέβαια ότι εκεί που υπάρχουν ήδη συνδέσεις ε, είναι πολύ σημαντικό να γίνεται και αντίστροφη ροή όταν υπάρχει το δίκτυο. Αυτό φάνηκε και το περασμένο Ιανουάριο, αλλά θα πρέπει να σκεφτούμε μήπως πρέπει να δημιουργήσουμε νέες εγκάρσιες συνδέσεις και αυτό αφορά εκείνους που είναι τελείως απομονωμένοι. Και αυτές οι χώρες είναι οι χώρες της Βαλτικής και η Φιλανδία, γιατί εξαρτώμαστε 100% από έναν προμηθευτή. Αντίστοιχα με την Ουκρανία, όπου τα προβλήματα ήταν μόνο πολιτικά κατά την άποψή μου. Ήτανε αποκλειστικά πολιτική απόφαση να σταματήσει, να κλείσει η στρόφιγγα. Αυτό μπορεί κάποια στιγμή να γίνει και στη δική μας περιοχή. Και ρωτώ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το έχει σκεφτεί αυτό και σε ποιο βαθμό. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Και τώρα η κυρία Κολάρσκα Βομπίνσκα. E, Ευχαριστώ πολύ. Ναι, χαίρομαι και εγώ πάρα πολύ που βλέπω την πρόταση αυτή να κατατίθεται. Αλλά τώρα μιλούμε για καταστάσεις έτσι, κρίσεων και πώς μπορούμε να τις προλάβουμε. Στο άρθρο 5 διαβάζουμε για ε, προληπτικά σχέδια δράσης που θα πρέπει λέει κάθε πέντε χρόνια να ε, ανανεώνονται όχι και κάθε πέντε χρόνια, κάθε χρόνο θα πρέπει και κάθε δύο χρόνια να ενημερώνονται εκτό των να θεωρούνται. Γιατί αν ξεσπάσει μια κρίση δεν μπορούμε να περιμένουμε δύο χρόνια για να προχωρήσουμε σε ένα ε, νέο σχέδιο ε, πρόληψης. Δεύτερο σχόλιο. Προηγουμένως κάποιος Ισπανός συνάδελφος εξήγησε πώς έχει κατάσταση στη χώρα του και είπε ότι είναι πολύ διαφορετική από ό,τι στις ανατολικές χώρες, τις χώρες της Ανατολικής Ευρώπης και θα πρέπει να ληφθεί υπόψη αυτό. Μα κατά την άποψή μου αυτό είναι αλληλεγγύη. Ότι είμαστε εδώ όλοι για έναν και ένας για όλους, ο καθένας για όλους. Δεν μπορούμε να έχουμε υπερβολικά ευέλικτη θεώρηση αυτών των θεμάτων. Ότι το α μας αφορά, το β δεν μας αφορά. Όπως είπε και ένας συνάδελφος προηγουμένως, συχνά ε, αυτές οι κριτικά κίνητρα. Γι' αυτό χρειάζεται και έχει τόσο μεγάλη σημασία η αλληλεγγύη, διότι ορισμένες χώρες βρίσκονται σε καλύτερη μοίρα από κάποιες άλλες. Ευχαριστώ η κυρία Νίμπλερ. Ευχαριστώ. Άργησα λίγο να έρθω και έχασα την παρουσίαση των εκπροσώπων της Κομισιόν και αν τυχόν επαναλάβω κάτι παρακαλώ να ε, συγχωρήσετε. Έχω ε, καταρχάς συγκεκριμένη ερώτηση και μετά παρατηρήσεις. Είναι γνωστές οι δομές της, ε, του φυσικού αερίου στα κράτη-μέλη υπάρχουν διαφορετικά γεωγραφικά δεδομένα και μία ε, πρόληψη και αντιμετώπιση της κρίσης διευκολύνεται πολύ περισσότερο όταν έχουμε ε, παρόμοιες προδιαγραφές και τεχνικά standards. Άρα λοιπόν πρέπει οπωσδήποτε να υπάρχει και ένα ποσοστό ευελιξίας για να μπορέσουμε να προσαρμοστούμε και ε, θα ήθελα να ρωτήσω γιατί ακολουθείτε την ε, νομοθετική πορεία ενός κανονισμού και όχι μιας οδηγίας δεδομένου ότι όπως είπαμε επισημείτε την ευελιξία στα κράτη-μέλη κάποια ε, ευελιξία χειρισμών ή κανονισμών γιατί δεν χρησιμοποιείτε μια οδηγία ως μέσον και όχι κανονισμό. Δεύτερη ερώτηση αφορά την κρίση του φυσικού αερίου τον Ιανουάριο Είχαμε λοιπόν την εμπειρία αυτή η οποία μας έδειξε ότι εάν οι εταιρείε συνεργαστούν και συντονιστούν το πρόβλημα μπορεί να λυθεί. Δεν λέω λύνεται αυτόματα αλλά είναι δυνατό να λυθεί. Και για την αντιμετώπιση της κρίσης θα πρέπει οι εταιρείε να αναλάβουν τις ευθύνες τους και θα πρέπει να δημιουργηθεί μία ταξινόμηση της, ευθύνη, της ευθύνης έτσι ώστε καταρχάς να την έχουν οι εταιρείε μετά το περιφερειακό ευρωπαϊκό επίπεδο και εν συνεχεία μία ανώτερη βαθμίδα ε, να κλιμακωθεί λοιπόν η ευθύνη έτσι ώστε και ιδιωτικοί φορείς ή εταιρείες ή δημόσιοι φορείς και εν τέλει ολόκληρη Ευρωπαϊκή Ένωση να μπορεί να γνωρίζει και να αναλαμβάνει τις συγκεκριμένε ευθύνε. Θα πρέπει, όπως είπα, επαναλαμβάνω, οι εταιρείε να αναλάβουν τις ευθύνε τους και πιστεύω και εγώ, όπως είπαν οι συνάδελφοι, ότι και τα κράτη-μέλη θα πρέπει αναλαμβάνονται τις ευθύνες τους να έχουν ένα μίνιμουμ προτύπων, μίνιμουμ από στάνταρτ τα οποία να εφαρμόζουν και μέσα στα πλαίσια της ε, αλληλεγγύης. Διότι η, το, η άλλη πλευρά του νομίσματος είναι να, μπορέσουμε να έχουμε ένα συντονισμό και μία αλληλεγγύη μεταξύ μας. Πολλές ερωτήσεις ε, και παρακαλώ να απαντήσει η Επιτροπή και έχετε και λίγο άνεση χρόνου. Ο κύριος Ρούτε, θα απαντήσω όσο μπορώ καλύτερα και ε, όταν δεν μπορώ άλλο θα δώσω το λόγο ή δεν ξέρω να απαντήσω, θα δώσω το, το λόγο στον συνάδελφό μου. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλα τα μέρη του Κοινοβουλίου για την πολύ θετική υποδοχή της ε, ε, πολύ θετική τους ε, αντιμετώπιση αυτής της ε, πρώτης συζήτησης και προσβλέπω με μεγάλη ικανοποίηση τις συζητήσεις που θα έχουμε τους επόμενους μήνες. Πιστεύω ότι θα μπορέσουμε να προχωρήσουμε γρήγορα σε αυτή την νομοθετική διαδικασία και πιστεύω ότι ο Επίτροπος Πίβαξ πιστεύει ακριβώς το ίδιο. συμφωνώ με τον εισηγητή για, για τον ορισμό του άρθρου 9 παράγραφος 6. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να ορίσουμε μια κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Προσπαθήσαμε να το κάνουμε αυτό στο άρθρο 9 σημείο 6, αλλά ακόμα χρήση βελτίωσης. Ε, θα το μελετήσουμε. Και ε, σύμφωνο επίσης ε, όταν θέλουμε να κάνουμε ένα fuel switching, αλλαγή καυσίμου δηλαδή, και να χρησιμοποιήσουμε, να χρησιμοποιηθεί ένα καύσιμο το οποίο είναι λιγότερο αποτελεσματικό σε σχέση με τις εκπομπές διοξιδίου, του άνθρακα, ε, όπως είχαμε αυτή τη συζήτηση και με την από ε, με, την, ε, με το κλείσιμο πυρηνικών εργαστησιών όταν λοιπόν κάνουμε αυτό το fuel ε, θα κοιτάξουμε και το θέμα του fuel switching για την ανταλλαγή πληροφοριών υπάρχουν πολλά πολλές και να, πολλές πρωτοβουλίες του τομέα αυτού, εμπορικές πρωτοβουλίες και μέσα στα πλαίσια του άρθρου 12.3 μπορούμε να εισαγάγουμε και, και, άλλες. Ήδη έχουμε ε, μία πρόβλεψη όσον αφορά την εμπιστευτικότητα ε, των πηγών, άρθρο 13, αλλά εάν θέλετε στη συζήτηση μπορούμε να ενισχύσουμε ε, την ε, διάταξη αυτή έτσι ώστε να ε, λαμβάνουμε τις πληροφορίες μόνο αυτές που χρειαζόμαστε έτσι ώστε να μην προκύπτει τόσο έντονο το θέμα της εμπιστευτικότητας. Όσον αφορά τον ορισμό του προστατευόμενου πελάτη, protective customer, εδώ ουσιαστικά στόχος μας είναι τα νοικοκυριά. Στόχος μας είναι να καλύψουμε τα νοικοκυριά και εν συνεχεία ας καθορίσουν τα κράτη-μέλη ε, ποιοι είναι οι άλλοι προστατευόμενοι ε, πελάτες, ε, μικρομεσαίες επιχειρήσεις, άλλοι φορείς. Αν και πρέπει να πω ότι ο προστατευόμενος πελάτης παίζει, έχει έναν ρόλο μόνο μέσα στο, στο πλαίσιο του ημέρου και του διμήνου. Μέσα σε αυτά τα πρότυπα, σε αυτά τα standards, όχι μέσα στο σύνολο της συνολικής, ε, των συνολικών αναγκών φυσικού αερίου, αλλά αυτών των δύο περιόδων, του ημέρου και των 60 ημερών. Αυτά λοιπόν για το προστατευόμενο πελάτη χάρηκα που άκουσα αρκετά μέλη να σχολιάζουν ε, πτυχές ε, πέραν του κανονισμού. Ο κύριος Ριτζίπ και ο κύριος Κάρενς και Μπαλτσίτης. που αναφέρθηκαν στην περιοχή της Βαλτικής και στις δυσκολίες εκεί. Συνεχίζουμε τις διαβουλεύσεις μας ή τις εργασίες μας μάλλον ε, στο ενεργειακό πρόγραμμα διασύνδεσης της περιοχής της Βαλτικής και στην στον ηλεκτρισμό αλλά και στο φυσικό αέριο και τις διασυνδέσεις του τομέα φυσικού αερίου. Διότι είναι αλληλένδετα, ε, αλληλένδετες οι ανάγκες ε, και στον τομέα του ηλεκτρικού, ηλεκτρισμού Θέλουμε βέβαια να διαχειριστούμε τον τομέα αυτό ώστε να μην υπάρχει υπερδυναμικό, πλεόνασμα δυναμικού όπως το έχουμε κάνει μεταξύ Σουηδίας και Λιθουανίας και θέλουμε να βρούμε και εναλλακτικέ λύσεις. Γι' αυτό θα χρειάζεται να εξετάσουμε ε, τις, ε, τις διασυνδέσεις φυσικού αερίου μεταξύ Λιθουανίας και Πολωνίας ποιος ε, όγκος ε, χρειάζεται, ε, επίσης τις διασυνδέσεις μεταξύ Φιλανδίας και Εσθονίας, η Λετωνία με τα αποθέματα της τι ρόλο παίζει, εμπορικές δηλαδή πτυχές τις οποίες πρέπει να εξετάσουμε. Όλα αυτά τα ερωτήματα απαντώνται καλύτερα σε περιφερειακό πλαίσιο και ο κανονισμός θα παρουσιάσει ακριβώς αυτό το πλαίσιο το περιφερειακό μέσα στο οποίο θα αναπτύξουμε τις δραστηριότητε μας ε, σε σχέση με τις βαλτικές διασυνδέσεις. Το, θέμα του προτύπου νη μείον για νέους για τις νέες καινούργιες ε, εταιρείες, καινούργιους ε, προμηθευτές, θα το εξετάσουμε θα το επανεξετάσουμε όσον αφορά την παροχή αδειών, τις αναγκαίες παροχές αδειών λειτουργίας νέων επιχειρήσεων προμηθευτών. Η κοινότητα υπό το άρθρο 10 κάνει μια, ένα πολύ λεπτό διαχωρισμό εάν ένα κράτος μόνο φύγεται μπορεί να κηρύξουμε κατά κατάσταση πρώτη ανάγκη. εάν όμως αφορά περισσότερο του ενός κράτη μέλη μπορεί να πούμε μια δεν θα κηρύξουμε γενικά κατάσταση έκτακτης ανάγκης αλλά ε, ενδέχεται να, να ενισχύσουμε στην περίπτωση αυτή τη συνεργασία μεταξύ των κρατών όταν υπάρχει κάποια διακοπή ή κάποια δυσχέρεια στην ροή του, του, του φυσικού αερίου. Κύριε Σμόποντα, νομίζω απάντησα στις περισσότερες ερωτήσεις. Και συμφωνώ μαζί σας ε, για την ασφάλεια του ε, φωδιασμού και της προμήθειας ενέργειας ότι δεν καλύπτεται μόνο από τον κανονισμό αυτό, είναι και ε, πολλά συμπληρωματικά στοιχεία. Θα ξανακοιτάξουμε τον ορισμό του N1. Θα πρέπει να ομολογήσω προς ντροπή μου ότι αν κοιτάξετε στο παράρτημα τον ορισμό του N 1, ούτε εγώ ο ίδιο δεν το καταλαβαίνω και χρειάζομαι να ρωτήσω και να ζητήσω τα φώτα των συναδέλφων μου για να μου τα εξηγήσουν. Νομίζω πραγματικά χωράει η διευκρίνηση εκεί. Ε, είναι σχεδόν μαθηματικός τύπος δηλαδή για να το καταλάβεις αυτή τη φόρμουλα των ήμιων 1 για τη δημοσίευση. Η επόμενη απάντηση κύριε Έντσου είναι σαφέστατο ότι θα πρέπει να εξασφαλίσουμε ε, πληροφόρηση ε, της Επιτροπής βάσει του άρθρου 12 να είναι η ε, κατάλληλη και πλήρης και ταυτόχρονα όμως να τηρείται και το απόρριτο και έχει μύθια στις περιπτώσεις αυτές όταν χρειάζονται προστασία. Κύριε Ντεάντζελης, με προκαλείτε. Να αρχίσουμε τώρα γενική συζήτηση για την ενεργειακή πολιτική. Γιατί ουσιαστικά ρωτάτε ακριβώς για το ενεργειακό μείγμα. Βεβαίως χρειαζόμαστε διαφοροποίηση των πηγών μας και των ε, οδών προμήθειας και των αγωγών, αλλά βεβαίως ε, επίσης χρειάζεται να δούμε και συνολικά το ενεργειακό μας μείγμα. Αυτό ξεπερνάει κατά πολύ τη βαρούσα ε, πρόταση κανονισμού που μας απασχολεί αυτή τη στιγμή. Με αυτά νομίζω απάντησα πάνω κάτω σε όλες τις ερωτήσεις. Αυτό που είπατε κυρία ε, Κολάρσκα Μπουλένσκα για την αναθεώρηση των ε, προγραμμάτων δράσης αναδιετία. Ε, συμφωνώ με αυτό που λέτε, αν υπάρχει κρίση δεν θα περιμένουμε δύο χρόνια για να αναθεωρήσουμε το πρόγραμμα. Κυρία Νίμπλερ. Νομίζω ότι προσπαθήσαμε κατά τη διάρκεια της συζήτησης σήμερα να ξεκαθαρίσουμε ε, μεγάλη σαφήνεια ότι είμαστε υπέρ του κανονισμού σε μεγάλο βαθμό που ε, βασίζεται κατά κύριο λόγο ε, στη δραστηριότητα των επιχειρήσεων. Κατά την άποψή μου μπορεί κανείς και με κανονισμό να βοηθήσει και να εφαρμόσει και την αρχή της επικουρικότητας όταν αφορά ο κανονισμός αυτό και οικονομικούς φορείς. Ε, λέμε κανονισμό για να προχωρήσουν τα πράγματα γρήγορα, να μην έχουμε τα προβλήματα που έχουμε τη μεταφορά ε, μιας οδηγίας που είχαμε στο παρελθόν και τα εξηγήσαμε στην έκθεσή μας όπου η εφαρμογή ήταν πάρα πολύ ε, κατακαιρματισμένη, ε, διαφορετική και σε μεγάλο βαθμό δεν εφαρμόστηκε καθόλου. Οπότε, ε, κανονισμός. Βεβαίως, σεβόμενοι πάντα την αρχή της επικουρικότητας και την πραγματικότητα σε κάθε κράτος μέλος. Κάθε χώρα ζει μια διαφορετική κατάσταση. Εξού και δεν έχουμε γενικές διατάξεις ή ενδείξεις ή υποδείξεις να έχει ο καθένας ε, απόθεμα χ, αλλά ε, μόνο ο κανόνας νη πλην ένα. Να μεταφερθεί αυτό στην εκάστοτε πραγματικότητα για την πρόληψη της κρίσης βασικά και μόνο σε τελική φάση και σε έκτακτη να δράει η Ευρωπαϊκή Ένωση όταν θα έχουν εξαντληθεί όλα τα επίπεδα και αποτύχει ξέρω εγώ, οι επιχειρήσεις, η τοπική αυτοδιοίκηση, τα κράτη τα λοιπά, να ε, ε, δράει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Νομίζω ότι τετραγωνίσαμε τον κύκλο τελικά. Ευχαριστώ. Ε, πολύ μεγάλη πληροφόρηση και ε, περισυλλογή και <laughs> Πολύ χαίρομαι πολύ. Το πιο ωραίο που άκουσα ήταν ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν καταλαβαίνει τα ίδια της τα κείμενα. Ένα ε, τυβό και την κακία μου. Δεν μπορούσα. Είπατε, εντάξει, μία φόρμουλα, έναν τύπο μαθηματικό δεν καταλαβαίνετε. Δεν μου άρεσε, <laughs> εν περιπτώσει. Λοιπόν, κυρίε και κύριοι, εξαντλήσαμε για σήμερα τη μερίσια διάταξη. Ραντεβού αύριο το πρωί για τη συνέχεια. σα ευχαριστώ πολύ και δεν πειράζει που τελειώνουμε. Δεν βλάπτει να τελειώνει κανείς καμιά φορά και νωρίτερα. Ευχαριστώ πολύ. Καλή σας επάνω. Τα λέμε αύριο το πρωί.